Επίσης, η προσχώρηση επιβεβαιώνει την ουσία της Ένωσης ως κοινότητα που βασίζεται στο δίκαιο με τις αξίες της νομικής βεβαιότητας. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης θα υπόκεινται στην ίδια εξωτερική παρακολούθηση και υποπτία των τάξεων τους, των αποφάσεών τους, όπως και τα κράτη-μέλη. Η προσχώρηση της Ένωσης στην ΕΣΔΑ συζητιέται επί 30 χρόνια περίπου και από πρακτικά και ουσιαστική, από πρακτική και ουσιαστική άποψη μπορούμε να πούμε ότι ο επίγον χαρακτήρας όλο και μειώνεται λόγω της πρόοδου της νομολογίας και των πρόσφατων εξελίξεων στην Ένωση. Αλλά στην πράξη το αντίθετο συμβαίνει. Υπάρχει επίγον χαρακτήρας ιδιαίτερα σήμερα για προκειμένου να γίνει αυτή η προσχώρηση. Γιατί? Διότι οι εξουσίε της Ένωσης επεκτάθηκαν και επεκτείνονται σε τομεί που αφορούν τα 27 κράτη-μέλη της Ένωσης. Άρα, οι πράξεις της Ένωσης πρέπει τα, οι πολίτες να έχουν δυνατότητα να έχουν πρόσβαση είτε μία πράξη παραβιάζει ανθρώπινα δικαιώματα, όπως εγγυάται η σύμβαση και, το, και τα πρωτόκολλα. Και αυτό έχουμε στη σχέση μεταξύ των δικαστηρίων Στρασβούργου και Λουσεμβούργου. Η κατάσταση δεν είναι τόσο πολύπλοκη όσο φαίνεται με μια πρώτη ματιά. Σε μεγάλο βαθμό αυτές οι σχέσεις είναι μια λειτουργία μεταξύ εξειδικευμένων δικαστηρίων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τον οποίων ο ρόλο είναι άσκηση εξωτερικού ελέγχου σχεδόν στι διεθνεί υποχρεώσει τη Ένωση λόγω τη προσχώρηση στην ΕΣΔΑ. Συνεπώ, η προσχώρηση δεν δίνει την, τις αρμοδιότητες που έχει το δικαστήριο του Λουξεμβούργου. Με την προσχώρηση η Ένωση απλώς γίνεται το 28ο μέλος της Σύμβασης και το Δικαστήριο του Λουξεμβούργου θα θεωρείται από το Δικαστήριο του Στρασβούργου ως εσωτερικό δικαστήριο. Όπως συμβαίνει με τις άλλες εθνικές συνιστώσεις. Με άλλα λόγια, η ΕΣΔΑ είναι ένα εργαλείο επικουρική προστασίας και τα ε, όργανα της Ένωσης με την προσχώρηση θα εξακολουθούν να έχουν την κύρια ευθύνη προκειμένου την τήρηση των δικαιωμάτων που είναι καταγραμμένα στο κόρπους αυτό. Από τη στιγμή λοιπόν που θα γίνει εσωτερικός Bill of Rights που περιορίζει τις εξουσίες των κοινωνικών οργάνων, ο μηχανισμός της ΕΣΔΑ θα πρέπει να το δούμε σαν έναν εξωτερικό περιορισμό στις, και έλεγχο στις δραστηριότητες της. Άρα την ευθύνη για την εσωτερική λειτουργία εξακολουθεί να έχει το δικαστήριο του Λουξεμβούργου. Το δικαστήριο του Στρασβούργου δεν είναι ανώτερο δικαστήριο. Δεν τίθεται θέμα ποιο δικαστήριο έχει τον πρωτεύοντα χαρακτήρα. Το δικαστήριο του Στρασβούργου απλώ θα προβλέπει του ελάχιστου κοινού παρονομαστέ που προβλέπουν οι εγγύησει τη ΕΣΔΑ και των πρωτοκόλων. Άρα η τεχνική φύση της σημερινή κατάστασης θα πρέπει να αποκατασταθεί. Αυτή τη στιγμή ένα θύμα, αν έχει εξελίξει όλα τα εθνικά και ε, ε, μέσα και μέσα της Ένωσης, θα πάει στο Σασβουργό, όχι κατά αυτού ο οποίος διέπραξε το αδίκημα κατά κάποιο τρόπο, αλλά κατά ενός περισσότερων κρατών μελών. Αν δια, διαπιστωθεί παραβίαση της ε, ΕΣΔΑ, δεν υπάρχει εγγύηση ότι η κατάσταση θα διορθωθεί υπέρ του θύματος, υπέρ του παθόντος μάλλον. Γι' αυτό χρειάζεται η προσχώρηση. Βέβαια, δεν έχω εντολή, ούτε με αρμόδιο. Είμαι μέλο τη κοινοβουλευτική συνέλευση και δεν μπορώ να ασχοληθώ με τι τεχνικέ λεπτομέρειε τη διαδικασία προσχώρηση. Αυτό θα γίνει σε διακυβερνητικό επίπεδο. Έχουμε λεπτομερή μελέτη για τα ε, νομικά και τεχνικά θέματα για την προσχώρηση από την Steering Committee, από την Οργανωτική Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με το τι προβλέπει αυτή η διαδικασία θα δοθεί στην Επιτροπή των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Κοινοβουλίου από τον Πρεσβευτή, δόθηκε μάλλον αυτά 22 Φεβρουαρίου. Για μας τους βουλευτές το σημαντικό είναι να μην βαλτώσουμε μέσα στις λεπτομέρειες. Εμείς θέλουμε να δοθεί ένα ισχυρό σινιάλο. Να αρχίσουν διαπραγματεύσεις σοβαρά. Να κρατηθεί η ορμή που έχει δημιουργηθεί. Οι διαπραγματεύσεις πρέπει να αρχίσουν ήδη τον Ιούλιο. Προσχώρηση της Ένωσης σε μια συνθήκη που έχει γίνει για τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης. Και τα 47 μέλη έχουν συλλογική ευθύνη με βάση την σύμβαση και αυτό θα πρέπει να συμπεριληφθεί στη διαδικασία προσχώρησης. Ας το αποφασίσουν οι εμπειρογνώμονες αν υπάρχει ανάγκη για ένα νέο, τροποποιητικό πρωτόκολλο ή αν ορισμένα θέματα μπορούν να καλυφθούν στην συνθήκη προσχώρησης ή αν και τα δύο είναι αναγκαία για να έχουμε γρήγορα θέση ενισχύ της ε, σύμβασης όπως προβλέπει το άρθρο 25 του 1969 ή αν θα χρησιμοποιηθεί ρήτρα opting out προκειμένου να ισχύσει όσο πιο σύντομα γίνεται η συμφωνία αυτή. Επίσης η προσχώρηση της Ένωσης στην ΕΣΔΑ σημαίνει προσχώρηση στο σύστημα της σύμβασης ως ορθώς λέγεται στην παραγραφό 5 δε, ορισμένα συμβούλια, ορισμένα σώματα συνδέονται με την σύμβαση. Το δικαστήριο του Στρασβού που εξασφαλίζει το σεβασμό της ε, σύμβασης, η κοινοβουλευτική συνέλευση η οποία αποφασίζει για τους δικαστές και το εποπτικό σώμα που, ε, που εποπτεύει την εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων. Η πρόσβαση τη ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει ότι χρειάζονται ορισμένε θεσμικέ μεταλλαγές στα θέματα αυτά. Παρά το γεγονός και μόλον τούτο ότι δεν έχω την εντολή να αναφερθώ στα θέματα τα οποία έχουν συζητηθεί εδώ, θα ήθελα να πω ορισμένα πράγματα σε σχέση με τον διορισμό, με την επιλογή των υποψηφίων και τον διορισμό των δικαστών. Οι δικαστέ εκλέγονται από την κοινοβουλευτική συνέλευση από ένα κατάλογο τριών υποψηφίων που υποφάλλονται από τα συμβαλώμενα μέρη στην σύμβαση, τα κράτη-μέλη ένας δικαστής ο οποίος έχει εκλεγεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, φυσικά θα έφερε και πρόσθετη εμπειρογνωμοσύνη στο σύστημα του Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο. Για να εξασφαλίσουμε ότι μόνο οι υποψήφοι του υψηλότερου δυνατού διαμετρήματος θα εκλεγούν, πρέπει οι εκλογές αυτές να είναι δίκαιες και διάφανες. Σε ορισμένε χώρες όπως το Βέλιο και την Λετωνία υπάρχει υπάρχει παρουσία των εθνικών αρχών. Στην, περίπτωση, στην επιλογή στη Σλοβενία εκλέγονται από τι εθνικέ κοινοβουλευτικέ αρχέ, Ο βαθμό στον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να ενδιαφερθεί για την εσωτερική διαδικασία διορισμού μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναπόκειται σε εσά. Είναι μια ευκαιρία όμω να φέρω στην προσοχή σας ένα σημαντικό ψήφισμα <clears throat> το 1646 του 2009 που ενεκρίθη από την κοινοβουλευτική μα συνέλευση το θέμα αυτό επί τη βάση μιας έκθεση που εξεπώνησε η Επιτροπή μας και που λέει ότι για την επιλογή των δικαστών το άρθρο 22 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης λέει ότι οι δικαστές επιλέγονται από κοινοβουλευτικές συνελεύσεις από ένα κατάλογο τριών υποψηφίων που αναφέρονται που επιλέγονται μάλλον από τις υψηλές συμβαλόμενες πλευρές. Επομένως με ενδιαφέρον αντιμετώπιζε την ιδέα που αναφέρεται στην παράγραφο 5 του να εξασφαλίσουμε τη συμμετοχή εκπροσώπων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην επιλογή δικαστών στο δικαστήριο του Στρασβούργου, στο ΕΔΑ. Κατανοώ ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να συζητηθεί και χωρισμένα από τις δύο κοινοβουλευτικές μας συνελεύσεις, παραλλήλως με την διαδικασία διαπραγματεύσεων προσχώρησης. Και κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου μια τελική παρατήρηση για το θαυμάσιο κείμενο του κυρίου Ραμών Χάουρεγη, κατά την άποψή μου η διατύπωση παραγράφου 6 φαίνεται ότι αποκλείει ε, προσφυγέ μεταξύ κρατών μελών με έναν τρόπο που είναι ιδιαίτερα ευρύ και διασταλτικός. Θα προέτεινα να διατυπωθεί, να αναδιατυπωθεί επί τη βάση του άρθρου 844 για τη συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να περιοριστεί σε διαμάχες που έχουν να κάνουν την εφαρμογή ή την ερμηνεία των συνθήκων. Τούτου λεχθέντος. Πρόκειται για ένα εσωτερικό θέμα που θα πρέπει να αποφασιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι φυσικά για την κυριολεκτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Επομένω, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας. Grazie lei per il suo intervento e adesso do la parola alla Ευχαριστούμε. Το λόγο η κυρία Φρανσουάζ Κούλκενς, Τούλκενς, δικαστής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Θα ακούσουμε με πολύ προσοχή τη μαρτυρία σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Επιτρέψτε μου να σα ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σα. Εγώ θεωρώ ότι είναι θαυμάσια αυτή η πρωτοβουλία να κάνετε μια ακρόαση για τα θέματα αυτά, γιατί νομίζω ότι αυτό θα μα επιτρέψει να διευκλευκάνουμε πολλά από τα ερωτήματα τα οποία θέτε εσεί στον εαυτό σα, αλλά και εμεί τον ίδιο ημών εαυτόν μα. Μπορεί κανεί να συζητήσει για τα πλεονεκτήματα τα οποία θα αποκομίσουν οι Ευρωπαίοι πολίτε για τα πλεονεκτήματα τη προχώρηση Για μένα, από την στιγμή που ετέθησε εφαρμογή η συνθήκη τη Λισαβόνα, αυτό το θέμα θεωρώ ότι έχει ουσιαστικά επιληθεί και όλα τα επιχειρήματα έχουν γίνει κατανοητά και περιλαμβάνονται στο σχέδιο εκθεσή σα, του οποίου τα συμπεράσματα συμμεριζόμαι απόλυτα. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, με την εφαρμογή τη συνθήκη τη Λισαβόνα, έχει ανοίξει ο δρόμο για την προσχώρηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση στη Σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ευκαιρία να συγκεκριμενοποιήσουμε αυτή τη δυνατότητα, η οποία πρέπει να ακολουθήσει δύο οδηγές αρχέ. Θα πρέπει το ταχύτερο δυνατό και με το πιο απλό δυνατό τρόπο να επιτευχθεί αυτή η συγκεκριμενοποίηση. Δεν σημαίνει αυτό θα είναι ταχεία και απλή η προσχώρηση. Προφανώ όχι και αυτό λόγω τη επαχθού και πολύπλοκη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 218 τη Συνθήκη για τη Λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά λόγω αυτή τη αυτή τη πολυπλοκότητα η οποία επιβάλλεται από τι συνθήκε, η δική μα απάντηση δεν θα πρέπει να είναι να προσθέσουμε και άλλα στοιχεία, αλλά θα έπρεπε να μειώσουμε στο ελάχιστο απαραίτητο τα στοιχεία αυτή τη σύμβαση, ώστε να μην καθυστερήσουμε αυτή την προσχώρηση για πολλά χρόνια, κάτι το οποίο θα ήταν λυπηρό. Και θα σα πω τώρα γιατί. Η ταχύτητα λοιπόν, το ταχύτητο δυνατό είναι η προσχώρηση. Γιατί? Γιατί υπάρχει το κατεπήγον. Εδώ και πολλά χρόνια το σύστημα τη σύμβαση αντιμετωπίζει μια έλλειψη ισορροπίας η οποία έχει και μια ένα χαρακτήρα ανομαλία. Ενώ όλα τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση υπόκειται στον εξωτερικό έλεγχο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ΕΔΑΤ, ακόμα και όταν εφαρμόζουν το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι αντικείμενο δικαίου. Και πρέπει να το τονίσω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να είναι διάδικο σε μια διαδικασία ενώπιον του ΕΔΑΔ, κάτι το οποίο μπορεί να οδηγήσει προφανώ προβλήματα για την εκτέλεση των αποφάσεων οι οποίε προκύπτουν από τη δικαστική διαδικασία όταν διαπιστώνεται μια παραβίαση της Σύμβασης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως στην περίπτωση της απόφασης Μάτιους. Και έχουμε υποσχεθεί στους πολίτες μας να ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα. Τώρα που είναι δυνατό να το κάνουμε, πρέπει να το κάνουμε με μεγάλη ταχύτητα και δεν θα πρέπει να χρόνο τριβήσουμε. Υπάρχει μια δεύτερη επιχειρηματολογία που κάνει σε αυτή την προσχώρηση με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Η χάρτα θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τονίστηκε αυτό πάρα πολύ σήμερα το πρωί, ότι είναι το πιο εξελιγμένο και το πιο σύγχρονο εργαλείο στον τομέα αυτό. Αυτή η χάρτα λοιπόν θεμελιωδών δικαιωμάτων ετέθη σε εφαρμογή. Γνωρίζουμε ότι αυτή η χάρτα περιλαμβάνει ένα μεγάλο μέρο των δικαιωμάτων που περιλαμβάνονται στη σύμβαση, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και προβλέπει τα δικαιώματα αυτά όπω θα ερμηνευτούν από το ΕΔΑΘ, θα πρέπει να είναι το ελάχιστο το οποίο θα πρέπει μέσα στο κοινοτικό δίκαιο. Σημαίνει αυτό σε πρακτικού όρου από την 1η Κεβρίου 2009 εναπόκειται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να εφαρμόσει και καταρχήν να ερμηνεύσει βάσει της χάρτας όλες τις διατάξεις οι οποίες είναι σημαντικές και ευαίσθητες σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Βέβαια, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει δώσει στο Δικαστήριο του Στρασβούργου σε τελική ανάλυση να εφαρμοσει και καταρχην να ερμηνευσει βασει τη χαρτα ολε τι διαταξει οι οποιε ειναι σημαντικε και ευαισθητε σε οτι αφορα την ευρωπαικη συμβαση ανθρωπινων δικαιωματων βεβαια η ευρωπαικη συμβαση ανθρωπινων δικαιωματων εχει δωσει στο δικαστηριο του στρασβουργου σε τελικη αναλυση να ερμηνευσει με αυθεντικό τρόπο τη σύμβαση αυτή χωρίς την παρέμβαση, χωρίς την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το δικαστήριο του Στρασβούργου δεν μπορεί να ασκήσει αυτή την ευθύνη σε σχέση με θέματα ερμηνείας της ε, σύμβασης αυτής από το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων όταν εφαρμόζει τη χάρτα ή σε υποθέσεις όπου είναι αρμόδια να αποφασίσει επί της ουσίας. Και εδώ είναι ένα κεντρικό σημείο. Τα δύο αυτά δικαστήρια του Λουξεμβούργου και του Στρασβούργου έχουν μια σημαντική αποστολή το κάθε δικαστήριο. Από τη μία πλευρά, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είναι ο εγγυητής της αυθεντικής εφαρμογής και ερμηνείας του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει την αποκλειστικότητα της ερμηνείας. Από την άλλη πλευρά, το ΕΔΑΔ είναι ο εγγυητής της ορθής εφαρμογής της, σύμβασης, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. <clears throat> Δεν μπορεί το ένα δικαστήριο ή το άλλο να υποκαταστήσει τα εθνικά δικαστήρια, ούτε το ΕΔΑΤ μπορεί να υποκαταστήσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σε σχέση με την εφαρμογή των συνθήκων. Επομένως, θα πρέπει να γίνει το ταχύτερο δυνατόν αυτή η προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο καλύτερος τρόπος είναι να το κάνουμε με ένα απλό τρόπο. Ο πιο απλός τρόπος δυνατός είναι και ο καλύτερος. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη. Η οδηγός αρχή μας θα πρέπει να είναι ότι μέσα στα πλαίσια της προσχώρησης αυτήν την σύμβαση η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να γίνει μια πλήρης συμβαλόμενη οντότητα σε αυτή τη σύμβαση, όπως και τα άλλα κράτη-μέλη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα γίνει τμήμα μιας ομάδος κρατών που συνδέονται μεταξύ τους με τα ίδια δικαιώματα και υποχρέωσεις στην εφαρμογή αυτής της σύμβασης και που είναι όλα ίσα ενώπιον της σύμβασης. Ο στόχος λοιπόν αυτής της προσχώρησης ήταν ακριβώς να υπόκειται η Ευρωπαϊκή Ένωση στον ίδιο εξωτερικό έλεγχο όπως και τα κρατη που την απαρτίζουν. Ένα υπερεθνικό λοιπόν έλεγχο. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα απολαμβάνει τον ίδιων δικαιωμάτων και θα υπόκειται στι ίδιε υποχρεώσει έναντι τη σύμβαση όπω τα κράτη-μέλη τη και ότι η έννοια τη ισότητα ενώπιον τη σύμβαση, που είναι μια ισχυρή έννοια, θα πρέπει να εφαρμόσει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βεβαίω η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι κράτο. Και θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη αυτό σε επίπεδο λειτουργία τη σύμβαση. Βάσει του πρωτοκόλλου 8 τη συνθήκη τη Λισαβόνα αναφέρεται και είναι λογικό εκπεφρασμένα ότι είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη οι ιδιαιτερότητες του ευρωπαϊκού δικαίου και στην περίπτωση αυτή είναι σαφέ ότι μια απόλυτη ισότητα μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Ένωση και των άλλων συμβαλωμένων κρατών μελών δεν είναι ούτε δυνατή ούτε επιθυμητή. Μόλον τούτο, μέσα στα πλαίσια τη προετοιμασία τη προσχώρηση θα πρέπει να μα οδηγήσει στο βαθμό του δυνατού η αρχή, η ισχυρή αυτή αρχή τη ισότητα ενώπιον τη σύμβαση και θα πρέπει να αποκλίνουμε από αυτή την αρχή μονάχα και μόνο στο βαθμό που αυτό είναι απαραίτητο για να σεβαστούμε την ιδιαιτερότητα και τον ειδικό χαρακτήρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και το δυνατόν περισσότερο το ίδιο καθεστώ που εφαρμόζεται στα κράτη-μέλη. Όχι μόνο γιατί αυτή είναι η πιο απλή λύση και γιατί είναι και ταχύτερη λύση, αλλά επίση και κυρίω κάτι που είναι πιο θεμελιώδη, γιατί δεν μπορούμε να δώσουμε την εντύπωση ότι μέσα στα πλαίσια του συστήματο τη Σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα υπάρχουν προνόμια των οποίων απολαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για μένα θα ήταν η χειρότερη υπηρεσία την οποία θα μπορούσαμε να δώσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αυτό θα υπέσκαπτε την αξιοπιστία τη, ενώ μέσω τη προσχώρησή τη προσπαθεί να επιτύχει ακριβώ το αντίθετο, να ενισχύσει αυτή την αξιοπιστία υποβάλλοντα τον εαυτό τη στου ίδιου εξωτερικού ελέγχου, όπω και τα κράτη-μέλη που την απαντήσουν. Ή κοθενοείται και επανέρχομαι, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τι ιδιαιτερότητε Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι πρόδειλο. Ακόμα και αν δεν το ζητούσε η συνδίκη τη Λισαβόνα, όπως φάνηκε και από μια τεχνική μελέτη που έγινε το 2000 στο Συμβουλίο της Ευρώπης σε σχέση με τι νομικέ και τεχνικές πτυχές της προσχώρηση και το οποίο είναι διαθέσιμο νομίζω σε αυτή την ακρόαση. Παραδείγματο χάρη, αναφέρθηκε και αυτό το θέμα σήμερα το πρωί από τον καθηγητή Ζακέ, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διαμοιράζεται ορισμένε αρμοδιότητε με τα κράτη-μέλη. Αυτό είναι μια σαφή ιδιαιτερότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία οπωσδήποτε πρέπει να ληφθεί υπόψη και εγώ συμφωνώ απόλυτα ότι δεν αναπόκειται στο δικό μα δικαστήριο να κρίνει για την κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και κρατών μελών. Και στο έγγραφο του 2002 υπήρχε αυτή η έννοια να είναι συνεναγόμενη η Ευρωπαϊκή Ένωση σε περιπτώσει κατά των κρατών μελών. Αυτή η πρόταση τώρα πρέπει να εξεταστεί σε βάθο. Και επομένω, θα πρέπει να την εξετάσουμε για να μπορούμε να βρούμε λύσεις οι οποίες θα μπορούν να οδηγήσουν σε ικανοποίηση όλων των εμπλεκομένων μερών. Γιατί το, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει κάποιες ιδιαιτερότητες που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Και αυτό αφορά επίσης και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Θα πρέπει να τροποποιήσουμε τη σύμβαση αυτή για να λάβει υπόψη τις ιδιαίτερες πτυχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά σεβόμενη την βαθύτερη φύση αυτή τη σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μεταξύ των σημείων τα οποία ήταν τα πιο σημαντικά στη συζήτηση του πρώην είναι αυτά που αφορούν τη δυνατότητα εσωτερικής προσφυγής. Για μένα θα πρέπει να αναλυθεί και θα πρέπει να εξεταστεί σε περισσότερο βάθος αυτή η ιδέα, αλλά με ένα καινούριο, με ένα νοπό πνεύμα. Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα αυτή, αυτό είναι ένα κεντρικό σημείο για το ΕΔΑΔ, θα πρέπει να είναι χρήσιμη τη διαδικασία, επομένως προσβάσιμη, αποτελεσματική και παρέχουσα ασφάλεια δικαίου. Και προφανώς η προδικαστική διαδικασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια διαδικασία η οποία εμφορείται από κοινή λογική, αλλά θα πρέπει να αναλυθεί. Οι αντιρρήσει που διατύπωσε ο δικαστή Τίμερσμαν σήμερα το πρωί θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και θα πρέπει να τι σκεφτούμε καλύτερα. Παρ' όλα αυτά, πρώτη απόψη <clears throat> είναι απαραίτητο να συζητήσουμε και πάλι αυτό το θέμα της εξάντλησης των ενδίκων μέσων προτού καταλήξουμε σε μια λύση, τουλάχιστον σε μια αναζήτηση λύσης σε ανώτερο επίπεδο. Και αυτή η ανάλυση θα πρέπει να έχει μερικά βασικά στοιχεία και νομίζω ότι εδώ συμφωνούμε απόλυτα, βρισκόμαστε στο ίδιο μήκο κύματο, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και το ΕΔΑΣ. Δεν θα πρέπει να ε, παραμελήσουμε τις πραγματικές <clears throat> αρμοδιότητες του κάθε δικαστηρίου. Θα πρέπει όλε οι σχέσει μα των δύο δικαστηρίων να γίνονται με αυτό το πλαίσιο. Δεύτερον, θα πρέπει να αξιολογήσουμε την σημασία τη κάθε κατάσταση όταν υπάρξει ένα δικαστήριο εθνικό το οποίο αρνείται να προβεί σε προδικαστική ερώτηση έναντι του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του Λουξεμβούργου. Θα ήταν λοιπόν ένα καλό μήνυμα να δώσουμε ότι αυτό είναι ένα σημαντικό σημείο. Ένα τρίτο στοιχείο το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι η χρονική προθεσμία. Όπω είπαμε σήμερα, δεν μπορούμε να υποχρεώσουμε τη δικαιοσύνη. Δεν είναι δυνατόν να, να ε, αποφασίσει μέσα σε ένα χρονικό διάστημα το οποίο δεν έχει όρια. Γι' αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντική η αρχή αυτή, μια θεμελιώδης αρχή και γι' αυτό αυτό το θέμα θα πρέπει να εξεταστεί ώστε να υπάρχει το ταχύτερο δυνατό μια λύση να μπορεί ένας ιδιώτης να ξέρει ότι η διαδικασία αυτή δεν θα οδηγήσει σε μια αυθαίρετη άρνηση του Εθνικού Δικαστηρίου να παραπέμψει μια ένα θέμα στι ελληνικέ καλένδε, παρα, μη παραπέμποντά το στο δικαστήριο του Λουξεμβούργου. Για μένα λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό οι διαπραγματεύσει οι οποίε θα γίνουν την προσχώρηση τη Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι ανοιχτέ διαδικασίε και επομένω εδώ υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα το οποίο θέλω να θίξω, δεν ξέρω πού ακριβώ βρίσκονται τα πράγματα αυτά. Το γεγονό ότι Ορισμένοι θέλουν να περιορίσουν την εντολή τη Κομισιόν Διαπραγματευτική στο πρωτογενέ δίκαιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν πράγματι όμω οι διαπραγματεύσει περιοριστούν μονάχα στο πρωτογενέ δίκαιο, αυτό είναι μια λανθασμένη προσέγγιση και θα οδηγήσει σε πάρα πολλού περιορισμού σε ό,τι αφορά τι διαπραγματεύσει. Για να κλείσω για ένα άλλο θέμα το οποίο ανέφερα προηγουμένως. Το βάρος εργασία στο Συμβούλιο. Προφανώς αυτό θα παίξει κάποιο ρόλο, διότι η προσχώρηση θα αυξήσει αυτό το βάρος. Ναι, πράγματι υπάρχει αυτό το άχρος, αλλά ξεκινήσαμε με ένα περιορισμένο χαρακτήρα ως δικαστήριο, γιατί σήμερα Υπάρχει όλο και περισσότερο έλεγχο των αποφάσεων που προκύπτουν μετά από μια προδικαστική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Δεύτερον, η προσχώρηση και το βάρος εργασίας είναι δύο προβλήματα τα οποία είναι διακριτά μεταξύ τους. Το <clears throat> πρωτόκολλο 14 θα τεθεί σε εφαρμογή στις 14, στην 1η Ιουνίου. Έχουμε ήδη την ε, συζήτηση και τη συμφωνία που έγινε στο Ιντελάκεν με στόχο να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα τη εφαρμογή αυτού του πρωτοκόλου όταν έχουμε ένα μεγάλο αριθμό προσφυγών. Ένα σημαντικό θέμα το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε και το θέμα τη επικουρικότητα. Τι σημαίνει επικουρικότητα, δεν σημαίνει ότι θα τα εγκαταλείπουμε όλα στα κράτη-μέλη, θα εξασφαλίσουμε αντίθετα ότι στα κράτη-μέλη υπάρχουν αποτελεσματικά ένδικα μέσα. Και τέλο, η προσχώρηση μπορεί να οδηγήσει και σε ένα ποιοτικό άλμα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα υπόκειται μονάχα στη σύμβαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα είναι και υπεύθυνη για την τήρησή του, αλλά θα μπορεί να παίξει και ένα ρόλο για την περαιτέρω ανάπτυξή τη. Αυτό μου φαίνεται ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Και τέλο, εφόσον μιλάμε για την προσχώρηση, δεν μπορούμε να δώσουμε εδώ πέρα μόνο την παράμετρο του βάρου εργασία. Η προσχώρηση θα οδηγήσει σε μια πιο συνεκτική κατάσταση, πιο σύμμορφη με τον τρόπο με τον οποίο οι θεσμοί μα σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, εξασφαλίζουν την ισότητα των κατορμενών σε ό,τι αφορά την ισότητα των πολιτών, σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή τη Ευρωπαϊκή Ένωση ω διάδικου σε διαδικασίε που την εμπλέκουν. Αυτά λοιπόν, κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρε, αυτοί είναι οι λόγοι για του οποίου, κατά την άποψή μου, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει το ταχύτερο δυνατό να γίνει μέλο τη Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Πρόκειται, σε τελική ανάλυση, για την διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ευρώπη, που είναι και το κοινό μα πληροδότημα. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία δικαστή Τούλκενς. Και το λόγο στον τρίτο εμπειρογνώμονα, τον κύριο Χριστόφερσεν που είναι εκτελεστικός διευθυντής του Ινστιτούτου Δανίας των Δικημάτων του Ανθρώπου. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε αξιότιμοι βουλευτές. Ε, στην παρούσα φάση είναι δύσκολο να προσθέσω πολλά στην συζήτηση που είναι ήδη πάρα πολύ επικοδομητική. Θα προσπαθήσω να ακολουθήσω την ε, δομή της έκθεσης ε, του εισηγητή σας, του κυρίου Ατόντου. Χαουρίς. Το Δανέζικο Ινστιτούτο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα είναι ένα εξάρτητο Ινστιτούτου έχουμε ένα μόνο θέμα στην ατζέντα μας, ανθρώπινα δικαιώματα. Και έχουμε ε, εντολή να παρέχουμε συμβουλές στην Δανέζικη κυβέρνηση και στο Δανικό Κοινοβούλιο και χαίρομαι που και εσείς το ίδιο ρόλο παίζετε από πλευράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δεν θα σας παρουσιάσω λοιπόν προσωπικές απόψεις για το θέμα, θα σας δώσω την επαγγελματική μου άποψη και θα προσπαθήσω να ε, διατηρήσω την αξιοπιστία μου χωρίς ε, να θέσω θέματα τα οποία μπορεί να είναι πολύ δύσκολα στην επίλυση. Θα ήθελα να πω ότι δεν θα αναφέρω όλες μου τις σημειώσεις, όλη μου την ομιλία. Μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε πάντως από το γραπτό κείμενο. Να περάσω σε ένα στοιχείο το οποίο θεωρώ ότι μπορεί να προσθέσει κάτι στην έκθεση. Μετά την παράγραφο ίσως ε, δύο θα μπορούσε να προσθεθεί ότι βάσει του πρωτοκόλλου 8 για την προσχώρηση αναφέρεται ότι σε ό,τι αφορά τις διευθετήσεις για την προσχώρια θα διασφαλιστούν τα διάφορα κριτήρια που αναφέρονται στα πρωτόκολλα. Άρα η Ένωση υποχρεούται να διασφαλίσει ότι τηρούνται όλα αυτά τα κριτήρια στις διαπραγματεύσεις για την προσχώρηση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ασφαλώς μπορεί να ψηφίσει και να αποφασίσει αν τηρούνται αυτά τα κριτήρια. Επίσης, χρήσιμο θα είναι να προσθέσουμε ίσως το εξή πριν από την παράγραφο 3 ένα καινούργιο στοιχείο την διατήρηση των ειδικών χαρακτηριστικών της Ένωσης και του κινητικού δικαίου, το οποίο δεν αναφέρεται ρητά στην έκθεση ως τώρα. Νομίζω ότι το ανέφερε η Επιτρόπος Ρέντινγκ, αποτελεί τμήμα της εντολής και είναι μια σημαντική αρχή γιατί θα πρέπει να συζητηθεί τι ακριβώς σημαίνει η έκφραση αυτή. Σημαίνει μόνο τις κοινέ αρμοδιότητες μεταξύ Ένωσης και κρατών μελών και τι σημαίνει ως προς τους μηχανισμούς αναθεώρησης. Πώς σχετίζεται με το στοιχείο αυτό, τι σημαίνει επίσης σε ό,τι αφορά τη φύση των δικαιωμάτων υπό τη χάρτα, ποια είναι η σχέση των δικαιωμάτων αυτών και των αρχών, των θεμελιδών αυτών δικαιωμάτων και πολλά άλλα θέματα τα οποία θα έπρεπε να συζητηθούν στον τομέα αυτών θα ανακύψουν. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό θα έπρεπε να προσταθεί στην έκθεση. Στην παράγραφο 3 τώρα γίνεται αναφορά στην ανάγκη να γίνει σεβαστή η κατάσταση των κρατών μελών σε ό,τι αφορά τις αποκλήσεις και τις επιφυλάξεις που έχουν διατυπώσει. Νομίζω ότι αυτό λίγο πολύ ανταποκρίνεται στο άρθρο 2 του πρωτοκόλου. Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι στην έκθεση αναφέρεται ότι οι επιφυλάξεις αυτές και οι αποκλήσεις δεν θα επηρεάσουν την νομική κατάσταση της Ένωσης σε ό,τι αφορά τη σύμβαση και ειλικρινά πιστεύω ότι εκεί θα ανακύψει το πιο σημαντικό πρόβλημα. Θα επανέλθω σε λίγα λεπτά στο θέμα αυτό, σχολιάζοντας την παράγραφο υπαριθμών 4. Να αναφέρω ένα θέμα το οποίο δεν έχουμε ακόμα συζητήσει σήμερα για τις αποκλήσεις. Πώς θα αντιμετωπίσουμε τις αποκλήσεις, αν υπάρχει κάποια απόκληση από την ε, Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Πώς θα επηρεάσει αυτό τις υποχρεώσεις των ε, κρατών μελών και τη σχέση των ε, κρατών μελών προς την Ένωση. Δεν έχουμε ακόμα τέτοιες απαντήσεις, δεν το έχουμε συζητήσει, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να το συζητήσουμε αυτό στις διαπραγματεύσεις τις επερχόμενες. στην παράγραφο 4. Είναι ένα, περιλαμβάνεται ένα από τα βασικά θέματα. Σε τι θα προσχωρήσει η Ένωση, στην Σύμβαση ή και στα πρωτόκολλα της Σύμβασης. Ακούσαμε να μιλάει η Επιτρόπος Ρέντινγκ για μια διπλή τακτική, διπλών, διπλό επίπεδο αν θέλετε και θα πρέπει η Ένωση να αποφασίζει από αυτού. Θα είναι μια δύσκολη απόφαση η οποία θα πρέπει να λεφθεί σε μετέπειτα χρονική στιγμή. Από πλευρά τη Ένωση είναι σαφέ ότι οι υποχρεώσει των κρατών μελών έναντι της σύμβαση δεν επηρεάζουν την προσχώρηση της Ένωσης στη σύμβαση. Αλλά γιατί λοιπόν αναφέρεται αυτό ω αρχή στο πρωτόκολλο. Ότι θα πρέπει να γίνουν σεβαστές οι θέσει των κρατών μελών και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι αποκλήσει και οι επιφυλάξει των κρατών μελών. Είναι δύσκολο το θέμα αυτό αν ένα κράτος ε, προσαχθεί στο Στρασβούργο σε περίπτωση επιφύλαξης ε, ή απόκληση σε περίπτωση που δεν έχει προσχωρήσει στο πρωτόκολλο. Η Ένωση μπορεί να ισχυριστεί ότι έχει πλήρη ε, νομική ευθύνη υπό τη σύμβαση. Αυτό μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα στο κράτος μέλος. και θα τεθεί θέμα αποδοχής ή όχι της ε, ε, δικαιοδοσίας του Στρασβούργου. Κάθε φορά που ένα κράτος μέλος δεν έχει πλήρη ευθύνη, η Ένωση δεν θα πρέπει να έχει πλήρες υποχρεώσεις. Αν αποδεχτούμε αυτή την ε, επιλεκτική προσέγγιση, τι θα σημαίνει αυτό για την προσχώρηση της Ένωσης. Θα σημαίνει ότι καταρχάς θα ε, γεμίσουμε χάσματα, τρύπες τουλάχιστον 10 κρατη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν επιφυλάξεις ή εξαιρέσεις, αν θέλετε, από τη Σύμβαση. Για το πρωτόκολλο 10, 10 κράτη-μέλη έχουν δηλώσει εξαιρέσεις και επιφυλάξεις. Για το πρωτόκολλο απαριθμών 4, 3 κράτη-μέλη έχουν επικυρώσει και 6 έχουν ε, επιφυλάξεις για το πρωτόκολλο υπερθμών 7. 3 κρατη κράτη-μέλη δεν έχουν επικυρώσει, δεν έχουν υπογράψει και 8 διατηρούν επιφυλάξεις για το πρωτόκολλο υπαριθμών 12. 20 κράτη-μέλη δεν έχουν υπογράψει ή επικυρώσει το πρωτόκολλο. Θεωρούμε λοιπόν ότι η ιδανική κυβέρνηση θα πρέπει να συνέλθει στο Στρασβούργο υπό το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να πει ότι όχι δεν μας δεσμεύει το πρωτόκολλο υπαριθμών 12 και η Ευρωπαϊκή Ένωση να πει ότι α, εμείς συμφωνούμε γιατί είναι το πρωτόκολλο υπαριθμών 12. Δεν νομίζω ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά ασφαλώς το Κοινοβούλιο θα πρέπει να ε, φροντίσει για μια ευρεία προσχώρηση. Λέμε στα Δανέζικα ότι έχει τρύπες σαν, ε, σαν ελβετικό τυρί. Αυτό θα γίνει και με την ε, προσχώρηση στη συνθήκη, αν επιλεχθεί αυτή η επιλεκτική μέθοδος ουσιαστικά. Για την παράγραφο 5 δεν θα επεκταθώ ιδιαίτερα. Πρόκειται για μια παράγραφο η οποία πραγματεύεται πιο τεχνικές πτυχές σε ό,τι αφορά την προσχώρηση. Θα ήθελα να αναφερθώ στην έκθεση της Διοικητικής Επιτροπής ε, της 28ης Ιουνίου 2002 του Συμβουλίου της Ευρώπης πριν από 8 χρόνια η Επιτροπή αυτή παρουσίασε τα πιο πολλά θέματα τα οποία θα πρέπει να εξετάσουμε από τεχνικής άποψης και συζητήσαμε κάποια από τα θέματα αυτά και σήμερα. Για την παραγράφη παραθυμόνα 6 μιλάμε για τις ε, διακρατικές ε, προσφυγές. Όπως είπε και ο δικαστής, Τούλκεν, η δικαστής δεν ε, είναι αυτός ο σκοπός να είναι ε, ενιαία και ισότιμη η συμμετοχή. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην μπορεί να προσαχθεί και αυτή σε μια τέτοια διακρατική ένσταση, αν θε προσφυγεί αν θέλει να έχει αξιοπιστία η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της προσχώρησης, θα πρέπει να αποδεχτεί αυτό το μηχανισμό διεθνούς ε, προσφυγής. Δεν θα πρέπει να κάνει opt-out, να αυτοεξαιρεθεί από αυτό το μηχανισμό. Πρόκειται για ένα πολύ κρίσιμο εργαλείο. Και θεωρητικά και στην πράξη σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Από πλευράς Ένωσης θα μπορούσε να πει κανείς βέβαια ότι είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικό ότι υπάρχουν χρονικοί περιορισμοί και δεν θα πρέπει να προσθεθούν νέε διαδικασίε με την Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Αλλά προφανώ και εμπλέκεται ένα νέο μηχανισμό για τι ευθύνε σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στην παράγραφο 7 αντιμετωπίζουμε το θέμα του ποιο θα πρέπει να είναι ο εναγόμενο σε περιπτώσεις ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για παραβίαση τη σύμβαση. Η βασική αρχή που πριτανεύει εδώ είναι ότι η αστική ευθύνη, η, ο τη αστική αστικής βασίζεται στο διεθνές δίκαιο, αλλά αλλιώ υπάρχουν τρει κατηγορίε που περιγράφονται επαρκώ πιστεύω στην έκθεση και φυσικά εξαρτάται από του ενάγοντε να αποφασίσουν εναντίον ποιου προσφεύγουν. Τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν τότε στη συνέχεια να αποφασίσουν ποιο έχει την ευθύνη και αυτό τελικά, σε τελική ανάλυση, θα πρέπει να διαλευκανθεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Λουξεμβούργου για το ποιο είναι υπόλογος βάσει του διεθνού δικαίου σε περιπτώσεις αυτού του είδους. όπω αναφέραμε προηγουμένω και στα πλαίσια του Οργανισμού Εθνών. Δεν είναι ένα ιδιαίτερο λοιπόν πρόβλημα σε πλαίσιο διεθνού δικαίου να αποφασίσουμε ποιο έχει την τελική ευθύνη. Αλλά κατανοώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει να αντιμετωπίσει ένα σημαντικό θέμα και θα έχει ίσω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση ιδέε για το πώ να αντιμετωπίσουν αυτό το θέμα που μπορούν να περιπλέξουν περισσότερο τα θέματα. Η διαδικασία συνε... συνεναγωμένης Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα στοιχείο πολυπλοκότητα το οποίο προστίθεται στο σύστημα. Αυτό αντιμετωπίζει στην παράγραφο 8 του το σύστημα αυτή τη στιγμή είναι ότι υπάρχει ένα εναγόμενο κράτος και οποιοδήποτε άλλο είναι τρίτος παρεμβαίνων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συμμετάσχει και πριν σαν τρίτος παρεμβαίνων σε διαδικασίες ενώπιον του ΕΔΑΔ και έχει λειτουργήσει αυτή η διαδικασία. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση ως τη αυτή δεν υπήρξε ποτέ διάδικος με στο σύστημα του ΕΔΑΔ. Αλλά μήπως θα έπρεπε να δεχτεί η Ένωση ότι είτε είναι τμήμα του συστήματος και πρέπει να αντιμετωπίζεται όπως οποιοδήποτε άλλος εναγόμενος, γιατί να έχουμε ένα ειδικό σύστημα, γιατί να εφεύρουμε μια νέα διαδικασία επειδή και μόνο πρόκειται για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί να υπάρχει ευνοϊκή και ειδική μεταχείριση για την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα στα πλαίσια της ΕΣΤΑ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αποδεχτεί τους κανόνες όπως έχουν και ας μην υπάρχουν ειδικέ ρυθμίσεις για αυτήν. σε γενικές γραμμές. Πιστεύω ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα θεωρείται υπόλογος για πολύ περισσότερες περιπτώσεις και τα κράτη-μέλη σε πολύ λιγότερες περιπτώσεις στο μέλλον. Έδωσε το παράδειγμα αυτό η Επιτρόπος Ρέντινγκ λέγοντας ότι αν ένα κράτος μπορεί να αποφύγει την ευθύνη βάσει της ΕΣΔΑ παραβιάζοντας το νόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τότε θα πρέπει να είναι συνεναγόμενη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι, δεν πρέπει να είναι συνεναγόμενη η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι ή εναγόμενη. Γιατί στην περίπτωση αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται πίσω από την παραβίαση από την πλευρά του κράτου τη ΕΣΔΑ, γιατί το κάνει αυτό το κράτο μέλο, γιατί δεν το εμποδίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκεί είναι λοιπόν το ερώτημα. Πρέπει να είναι η, το κράτο μέλο ή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ήταν και το αντικείμενο τη περίπτωση Μπόσφορου κατά τη Ιρλανδία. Και πρέπει να αποφασιστεί ποια θα είναι η πραγματικότητα σε αυτή την περίπτωση αλλά ίσως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αποκτήσει ένα μεγαλύτερο ρόλο από ό,τι προβλέπεται στην τωρινή έκθεση. Είναι ένα δύσκολο θέμα και νομίζω ότι είναι ένα από τα πράγματα τα οποία θα περιπλέξουν ακόμα περισσότερο τι διαπραγματεύσει ένταξη τη Ευρωπαϊκή Ένωση και δικαίω. Επίση, θα ήταν επιθυμητό, πιστεύω, η έκθεση να περιλάβει ένα τμήμα για το δικαίωμα να υπάρχουν αποτελεσματικές θεραπείες μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας. Αυτό θα μπορούσε να είναι κάπου μετά την παράγραφο 8. Συζητήσαμε το θέμα, όπως είπε η κυρία Τούλκενς, πρέπει να το εξετάσουμε ενδελεχώς. Ο κύριος Τιν, Τίμερμανς έκανε κάποιες παρατηρήσεις για το θέμα αυτό λέγοντας ότι είναι πάρα πολύ πολύπλοκο το πρόβλημα αυτό, αλλά γενικά δεν μπορούμε να ζητήσουμε από τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να, να εξαντλήσουν ε, εσωτερικά ένδικα μέσα, εάν δεν υπάρχουν αυτά τα εσωτερικά ένδικα μέσα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε αποτελεσματική θεραπεία σε όλες τις περιπτώσεις του ευρωπαϊκού δικαίου. Αυτό διεφάνηκε στην περίπτωση Μπόσπορους όταν είπε το δικαστήριο το σύστημα αυτό είναι συγκρίσιμο αλλά όχι ισοδύναμο. Και πιστεύω ότι πολύ εύκολα μπορείτε να βρείτε περιοχές δικαίου όπου δεν έχουν τα άτομα αποτελεσματικά ένδικα μέσα κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γιατί γίνεται αυτό, γιατί η βασική μνήα που υπάρχει στο σύστημα δεν είναι μια αποτελεσματική θεραπεία υπέρ των μεμονωμένων διαδίκων, είναι μια διαδικασία για συνεργασία των δικαστηρίων. Επομένω δεν μπορούμε να ζητήσουμε από του πολίτε από του μεμονωμένου διαδικού να καταφέρουν σε διαδικασίε οι οποίε δεν έχουν αποτελεσματικό χαρακτήρα. Ίσως κάτι το οποίο θα ήταν μια ενδιάμεση λύση, η οποία μπορεί να γίνει χωρίς μεγάλες δυσκολίες, είναι το δικαστήριο του Λουξεμβούργου, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, να πει ότι εμείς παροτρύνουμε τα κράτη-μέλη, τα δικαστήρια των κρατών μελών, να ζητούν να υπάρχει προδικαστικό ερώτημα εάν υπάρχει ένα πραγματικά ουσιαστικό θέμα θεμελιωδών δικαιωμάτων. Τότε θα μπορούσαν να κάνουν προδικαστικό ερώτημα τα εθνικά δικαστήρια και να υπάρχουν πολύ περισσότερες περιπτώσεις στο δικαστήριο του Λουξεμβούργου που φτάσουν στο Στρασβούργο. Και αυτό θα μπορούσε να γίνει χωρίς να τροποποιηθεί η συνδική της Λισαβόνας που πολλοί από εμάς θεωρούν ότι δεν είναι η κατάλληλη λύση για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα αυτά. Είμαι άχρονος, έχω ξεπεράσει το χρόνο μου, αλλά θέλω να κάνω μια παρατήρηση σε κάτι το οποίο ελέγχθη προηγουμένως από τον κύριο Μέσσερ Σμιτ και κάποιον άλλο μιλητή, πώς αντιμετωπίζουμε περιπτώσεις συγκρουωμένων δικαίων ποια είναι τα δικαιώματα, τα, τα, δικαιώματα τα οποία υπερέχουν όταν συγκρούεται η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με τη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και εγώ συμφωνώ με την αντίληψη ότι πρέπει να είναι αυτά τα οποία παρέχουν την καλύτερη προστασία. Φυσικά πρέπει να επιλύσουμε τη διαμάχη μεταξύ αυτών των δικαιωμάτων και πιστεύω ότι η ευρωπαϊκή πλευρά, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουν να πούνε ότι θα είναι αρμόδιο το δικαστήριο του Λουξεμβούργου, ενώ αυτοί που υποστηρίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα θα αποτιμούσαν να είναι το Στρασβούργο. Και εγώ, επειδή είμαι τη τελευταία άποψη, θεωρώ ότι πρέπει να είναι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Στρασβούργου πρέπει να έχει τον τελικό λόγο βάσει τη Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αυτοί πρέπει να κάνουν την τελική εξισορρόπηση δικαιωμάτων και συνέβη προηγουμένω και στην περίπτωση Φαν Hanover που αφορούσε την ε, ιδιωτικότητα και την ελευθερία έκφρασης και αποφασίστηκε κάτι από το Γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο, αλλά το Στρασβούργο ανέτρεψε αυτή την απόφαση. Μπορεί ο καθένα να έχει τη δική του ερμηνεία για τα θέματα αυτά. Οι έξυπνοι άνθρωποι γενικά έχουν αποκλίνουσε απόψει, αλλά τελικά ο τελικό θεματοφύλακα είναι το δικαστήριο του Στρασβούργου. Αυτή είναι η απόψή μου και από ό,τι κατάλαβα, από ό,τι είπε και ο Γερμανό συναδελφό μου, έχει ενσωματωθεί στο γερμανικό σύστημα αυτή η λύση και αυτό είναι ένα ιστορικό ορόσημο σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο στόχος μας είναι να κάνουμε πιο απλό το σύστημα λοιπόν, να αντιμετωπίσουμε τα θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να μην περιπλέξουμε πολύ τα πράγματα, γιατί μπορούμε να φτάσουμε σε ένα επίπεδο μεγάλης πολυδεδαλότητος. Ελπίζω ότι αυτά θα μπορέσουν να λειτουργήσουν μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια Το κείμενο της Κομισιόν στο δανεικό δελτίο ενημέρωση είπε ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον πέντε χρόνια, ελπίζω να γίνει νωρίτερα πάντως. Grazie. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Μπορούμε να ξεκινήσουμε τώρα τη συζήτηση για διάλογο. Έχουν οι συνάδελφοι τη δυνατότητα να λάβουν το λόγο, φυσικά και οι εμπειρογνώμονες εφόσον θέλουν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχάς, μια γρήγορη ερώτηση, η οποία νομίζω ότι μπορεί να απαντηθεί και εξίσου γρήγορα. Και μετά να κάνω και μια δήλωση. Αναφέρθηκε ότι κάποια κράτη-μέλη της ε, του Συμβουλίου της Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν έχουν υπογράψει ή έχουν εκφράσει επιφυλάξεις για τα πρωτόκολλα της Σύμβασης. Σήμερα το πρωί, από αυτά που μας είπε η Επιτροπός Ρέντινγκ, καταλάβαμε ότι δεν έχει αποφασιστεί ακόμα ποια πρωτόκολλα, σε ποια πρωτόκολλα θα προσχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ερωτώ λοιπόν, αν η Ευρωπαϊκή Ένωση προσχωρήσει σε ένα πρωτόκολλο, τα κράτη-μέλη και ένα κράτος μέλος δεν έχει προσχωρήσει στο πρωτόκολλο αυτό. Το πρωτόκολλο αυτό φαντάζομαι ότι θα καταστεί τμήμα του κοινωτικού δικαίου και θα πρέπει να εφαρμοστεί στο κράτος μέλος παρά τη θέληση της κυβέρνησης που αρνήθηκε να το υπογράψει και μια δήλωση, μια παρατήρηση για το τελευταίο που ανέφερε ο κύριος Κριστόφερσεν. Τι θα συμβεί αν υπάρχει δύο, σύγκρουση δύο δικαιωμάτων. Είπε ο κύριος Κριστόφερσεν ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε ποιο δικαίωμα δικαστηρίου θα προηγηθεί. Νομίζω ότι πιο σημαντικό είναι να κοιτάξουμε το σημαντικό ερώτημα του πού σταματάει το ένα δικαίωμα και πού αρχίζει το άλλο, αν υπάρχουν δύο συγκρουόμενα δικαιώματα, για παράδειγμα το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης και αφετέρου το δικαίωμα της ανεξιθρησκείας. Τι θα συμβεί και πώς μπορούμε να επιτρέψουμε να υπάρξουν παράλληλα και τα δύο αυτά τα δικαιώματα σε ό,τι αφορά τέτοια αντικρουόμενα συμφέροντα και δικαιώματα. Δεν θα ήταν καλύτερα αν το Συμβούλιο της Ευρώπης κάτσει και ξαναγράψει πού σταματάει η ελευθερία της έκφρασης και πού ξεκινούν τα υπόλοιπα δικαιώματα, προκειμένου να μην υπάρχουν αμφιβολίες, για να μην βρίσκονται σε μια τέτοια ενδιάμεση κατάσταση τα δικαστήρια και να πρέπει να αποφασίζουν αναπερίπτωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ως Εγώ θα ήθελα να έχω την άποψη του εκπροσώπου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που ήταν παρόν και στο πρώτο τμήμα του απογεύματος και να το θέσω δύο ερωτήματα τα οποία μου φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ απαραίτητο να τεθούν. Έχει το Συμβούλιο της Ευρώπης κάποια πρόθεση να δημιουργήσει ένα, ένα οργανισμό διαπραγματευτικού χαρακτήρα ad hoc. Ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλά ψηφίσματα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης σε σχέση με την ανάγκη να υπάρξει η προσχώρηση της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα υπάρξει κάποιος φορέας που θα αναλάβει τις διαπραγματεύσεις από την πλευρά του Συμβουλίου της Ευρώπης, η Επιτροπή Υπουργών, ίσως κάποια αντιπροσωπή από τη Γραμματεία του Συμβουλίου. Ποιος θα το επομιστεί αυτό. Δεύτερο ερώτημα, το οποίο για μένα είναι επίσης πολύ σημαντικό, είναι το εξή. Αποκτά περισσότερη αποδοχή η ιδέα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συμμετέχει στην επιλογή των δικαστών. Το λέω αυτό γιατί το ερώτημα είναι αν είναι δυνατό να γίνει αυτό σε μια κοινοβουλευτική συνέλευση που ήδη έχει κανόνες λειτουργίας. Πώς μπορούν να τροποποιηθούν αυτοί οι κανόνες μεταξύ των οποίων η ίδια η σύνθεση της κοινοβουλευτικής συνέλευσης. Κάποια μέρα πρέπει να αλλάξουν αυτοί οι κανόνες ώστε να είναι δυνατόν να υπάρχουν κάποιοι εκπρόσωποι οι οποίοι προέρχονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Πουχού και οι οποίοι εκείνη τη συγκεκριμένη ημέρα θα πρέπει να συμμετάσχουν στην κοινοβουλευτική συνέλευση η οποία ήδη έχει μια συγκεκριμένη σύνδεση. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω πώς θα γίνει. Θα μου φαινόταν πολύ απλούστερο η Ευρωπαϊκή Ένωση να στείλει τις υποψηφιότητες που θέλει να υποστηρίξει για, δικαστη... για δικαστές και μετά να εκλεγούν όλοι αυτοί από την κοινοβουλευτική συνέλευση. Να μην υπάρξει μια αγνήσια εκπροσώπηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην κοινοβουλευτική συνέλευση αλλά ξέρω ότι στην διαπραγματευτική της εντολή η Κομισιόν περιλαμβάνει και αυτή την ιδέα να υπάρχουν εκλογέ από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήθελα να ρωτήσω πώ θα γίνει αυτό το πράγμα στην πραγματικότητα. Ένα ακόμα ερώτημα σε σχέση με τον κύριο Κριστόφεσον, σε αυτά που είπε σε σχέση με το ρόλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση ω συνεναγόμενη. Πολύ καλό είναι να θέλουμε να πλησιάσουμε στο δυνατό την κατάσταση ενός κράτους, το οποίο είναι συμβαλόμενο σε αυτή την σύμβαση. Μπορούμε να το κάνουμε, αλλά δεν είναι σωστό αυτό απόλυτα, γιατί δεν είναι το ίδιο πράγμα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν νομίζω ότι μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να συμμετέχει, να ζητά να συμμετέχει σε όλες τις περιπτώσεις που τίθεται να αμφιβόλο το ευρωπαϊκό δικαίο, δεδομένου τα κάτι μέλη σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του κοινωτικού δικαίου, που λαμβάνουν ενός ευρύτατου ε, περιθωρίου εκτίμησης. Αν βάλουμε λοιπόν, το, αν θέσουμε το παράδειγμα μιας οδηγίας που τα κράτη-μέλη ένα κράτο μέλο ενάγεται γιατί εφάρμοσε με το δικό του, με το τρόπο μία οδηγία, τότε δεν ξέρω κατά πόσο θα πρέπει να υπάρχει επιπλέον και η παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να υπερασπιστεί το κοινοτικό δικαίωμα. Γιατί πρέπει λοιπόν να μην έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση το δικαίωμα υποστήριξης του δικού του κοινοτικού δικαίου όταν αυτό τίθεται ένα αμφιβόλο. Δηλαδή όταν έχει ένα κράτος μέλος ένα περιθώριο εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου, το οποίο είναι πάρα πολύ ευρύ, γιατί να μην μπορεί να υπερασπιστεί η Ένωση το κοινοτικό δίκαιο. Ευχαριστώ κύριε Χαουρέγγι. Ο κύριος Νταφ έχει το λόγο. Ε, ε, ε, Πρόεδρε, δύο ερωτήσεις έχω να θέσω. Προσπαθώντας να προκαταβάλουμε, αν θέλετε, και να προβλέψουμε πόσο θα δύσκολη θα είναι η προσχώρηση σε οποιοδήποτε σύμβαση, θα μπορούσε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου, ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Ευρώπης, να μας εξηγήσει το δύσκολο και περίπλοκο πλαίσιο το οποίο δημιουργείται από την θέση εφαρμογή του πρωτοκόλλου υπαριθμών 14. Μας κάνει εντύπωση το γεγονός ότι η συνθήκη αυτή θα πρέπει να περάσει από 74 εθνικά κοινοβούλια. Από 47 εθνικά κοινοβούλια. Προκειμένου να για να επικυρωθεί η πλευρά από, τη, από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν θέλετε, το πρωτόκολλο. Δεν θα είναι εύκολο. Αυτή είναι η εμπειρία που είχε το Συμβούλιο Μάλλον θα ήταν χρήσιμο να ακούσουμε την εμπειρία του Συμβουλίου της Ευρώπης ε, από τις ε, προηγούμενες επικυρώσεις. Κατά δεύτερον, όπως ξέρετε, υπάρχουν ασυνέπειες μεταξύ της Χάρτας των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων σε ό,τι αφορά το ΕΔΑΔ, σε ό,τι αφορά το πεδίο εφαρμογή. θεωρείτε ότι μακροπρόθεσμα όσο αναπτύσσεται στο Λουξεμβούργο ε, μεγαλύτερη δικαιονομολογία βάσει της ερμηνείας ε, της χάρτας μακροπρόθεσμα θα μειωθεί σε σημασία, θα υποσυνομευτεί το σύστημα του ΕΔΑΤ. Η προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύμβαση θα δώσει μεγαλύτερες δυνατότητες για την υπονόμευση του συστήματος του ΕΔΑΔ ή θα το ενισχύσει. Καταλαβαίνω ότι είναι αρκετά υποθετική ερώτηση αυτή. Και ίσως να μην απασχολεί άμεσα σε ό,τι αφορά τη διαπραγμάτευση της συνθήκες, αλλά θα με ενδιέφερε να ακούσω ποια είναι η γνώμη των εμπειρογνωμόνων από αυτού. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κυρία Γκάλ. Θα σταθώ στο ερώτημα το οποίο έτεθη ήδη από τον εισηγητή, γιατί πιστεύω και συμμερίζομαι τις ανησυχίες του. Ξέρω ότι είναι προβληματικό και δύσκολο το πώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα εμπλακεί στη διαδικασία επιλογής των δικαστών του ΕΔΑΔ. Είναι εφικτό λοιπόν, είναι δυνατόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να, να εκλέγει δικαστές οι οποίοι προστίθενται σε αυτούς της κοινοβουλευτική συνέλευση. Αυτό είναι το ερώτημα το οποίο εγώ θα ήθελα να προσθέσω στα προηγούμενα ερωτήματα. Ευχαριστώ. Δίνω τώρα το λόγο στους εμπειρογνώμονές μας για να δώσουν τις απαντήσεις τους, εάν θέλουν να απαντήσουν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να απαντήσω στο ερώτημα που αφορά τη διαδικασία εκλογής των δικαστών και επίσης αυτό που αφορά τη γενική κατάσταση της Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και το μέλλον το οποίο μπορούμε να ατενίσουμε. Νομίζω ότι εδώ ο εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου θα αναφερθεί στο θέμα αυτό για την διαδικασία επιλογής και εκλογής των δικαστών. Πρώτα απ' όλα θέλω να αναφέρω για μια ακόμα φορά ότι θα ήθελα να, δώσω στο, να ζητήσω από τον πρόεδρο τη δυνατότητα να διανεμηθεί το έγγραφο αυτό από την κοινοβουλευτική μα συνέλευση, το οποίο ανέφερα προηγουμένως. Και είναι ένα έγγραφο πληροφορικό από την ε, συνέλευσή μας για την Υποεπιτροπή Επιλογής Δικαστών που αφορά τη διαδικασία επιλογής των δικαστών του ΕΔΑΔ. Είναι σαφές από το έγγραφο αυτό που περιέχει λεπτομερεί πληροφορίες πώς γίνεται αυτή η διαδικασία. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε επέκεινα αυτά, αυτόν που ορίζει το άρθρο 22 της Σύμβασης που λέει ότι υπάρχει μία συγκεκριμένη διαδικασία βάσει της οποίας κάθε υψηλή συμβαλόμενη πλευρά θα πρέπει να παρουσιάσει ένα κατάλογο υποψηφίων τριών τον αριθμό που θα πρέπει να υποδειχθούν από τα υψηλά συμβαλόμενα μέρη. Αυτό σημαίνει ότι με τη διαδικασία προσχώρηση θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να παρουσιάσει και αυτοί τρει υποψηφίου. Αυτό είναι η προπόθεση για τη διαδικασία και αυτό είναι μια απέτηση η οποία δεν μπορεί να τροποποιηθεί γιατί αυτό περιλαμβάνεται στο κείμενο τη σύμβαση. Για όλα τα άλλα τα υπόλοιπα προσπάθησα να το εξηγήσω στο παρελθόν διάφορε φορέ και αντανακλάται σε μεγάλο βαθμό στο περιεχόμενο της παραγράφου 5 της έκθεσης του κ. Χαουραγή που θίγει ορισμένα θέματα τα οποία θα πρέπει να τύχουν ε, διασαφήνιση και διαπραγμάτευση μεταξύ των δύο πλευρών, μεταξύ της κοινοβουλευτική Συνέλευσης αφενός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αφετέρου. Πουχού τονίστηκε αυτό προηγουμένω ότι θα πρέπει τα δύο κοινοβουλευτικά σώματα να διαπραγματευθούν παράλληλα με τις διαπραγματεύσεις προσχώρησης την διαδικασία αυτή. Γιατί είναι απαραίτητο αυτό. Είναι απαραίτητο γιατί η Υποεπιτροπή για το Διασμό των Δικαστών στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης συγκροτείται σε διάφορα επίπεδα. Απαρτίζεται καταρχήν από τους εκπροσώπους που υποδεικνύονται από τις πολιτικές ομάδες, αλλά όχι από τα κράτη-μέλη της Σύμβασης. Γι' αυτό το λόγο το 47 μέλλον. Γι' αυτό υπογραμμίζω την συμμετοχή των υψηλών συμβαλωμένων μερών, διότι σε αυτή την περίπτωση ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι καλόδεκτος γιατί εμπλέκονται μεν πολλά εθνικά κοινοβούλια σε αυτή τη διαδικασία, αλλά η εμβέλεια της συμμετοχής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι κάτι το οποίο εναπόκειται σε εσά καταρχήν να το αποφασίσετε και μετά να το διαπραγματευτείτε με την Κοινοβουλευτική Συνέλευση Συμβουλίου τη Ευρώπη, ή να το συζητήσετε μέσα στι ομάδε εργασία. Γιατί χρειάζεται να θεσπιστούν σαφείς κανόνες ε, για να καθορίσουμε σε ποιο βαθμό τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα μπορούσαν να συμμετάσχουν στην υποεπιτροπή επιλογής των δικαστών για το ΕΔΑΔ, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι υψηλές συμβαλόμενες πλευρές είναι αυτές οι οποίες έχουν το δικαίωμα παρουσίασης υποψηφίων όπως είναι η πάγια πρακτική στο Συμβουλίο της Ευρώπης. Και αυτή είναι η βάση με την οποία λειτουργεί η Υποεπιτροπή επιλογή Δικαστικών. Σε ό,τι αφορά περαιτέρω την πρόταση για το δικαίωμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να έχει εκπροσώπους μέσα στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση για το σκοπό της ψηφοφορίας. Και αυτό είναι θέμα συζήτησης για διαπραγμάτευση μεταξύ των δύο κοινοβουλευτικών φορέων πιστεύω το σημαντικό είναι να ξεκινήσουμε τη συζήτηση, γιατί υπάρχουν ορισμένα θέματα τα οποία είναι σαφή και δεν απαιτούν ιδιαίτερη συζήτηση. Το γεγονός δηλαδή ότι τα υψηλά συμβαλόμενα μέρη θα πρέπει να είναι παρόντα και να έχουν το δικαίωμα να παρουσιάσουν ένα κατάλογο υποψηφίων, αλλά τελικά το τι θα πράξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εναπόκειται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να το προτείνει και να το διαπραγματευτεί με την Κοινοβουλευτική Συνέλευση και επίσης είναι γεγονό ότι μπορούμε να αλλάξουμε του κανόνες που προκύπτουν από τη Σύμβαση ότι ο κάθε δικαστή εκλέγεται από την Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου τη Ευρώπη. Μετά από όλα αυτά, η κατάσταση είναι σαφής, γιατί όλα αυτά είναι περιεχόμενο τη ΕΣΔΑ, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Για μία λοιπόν φορά και πάλι, ξαναεπαναλαμβάνουν, θα ήθελα να σας δώσω αυτό το μήνυμα. Ο βαθμός στον οποίο εσείς θέλετε να συμμετάσχετε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε αυτή τη διαδικασία εναπόκειται σε εσά τους ιδίους. Και στη συνέχεια θα πρέπει να υπάρξει διαπραγμάτευση μεταξύ των δύο κοινοβουλευτικών φορέων, ώστε να συζητηθεί και να επιληθεί το θέμα αυτό με την δημιουργία σαφών κανόνων, διαδικασίες που θα πρέπει να ή να συνάδει και με τις απαιτήσει της ΕΣΔΑ. Ο κύριος ε, κύριε Τούλκενς. Χωρίς μικρόφωνο κυρία Τούλκενς. Μικρόφωνο. Συγγνώμη, εδώ δεν έχω καμία απολύτως αρμοδιότητα για να αναφερθώ στο θέμα της εκλογής των δικαστών. Το ουσιαστικό είναι να υπάρχουν δικαστέ οι οποίοι αντανακλούν τι αξίε και τι αρχέ Ευρωπαϊκή Ένωση και τη δικαστική του κουλτούρα. Οποιαδήποτε διαδικασία λοιπόν η οποία θα εξασφαλίσει ότι οι δικαστέ αυτοί θα εξασφαλίζουν αυτέ τι ιδιότητε είναι πάρα πολύ σημαντική. Αλλά εγώ θέλω να λάβω το λόγο σε ένα άλλο θέμα που βρισκόταν μέσα στα πλαίσια τη προηγούμενη ερώτηση που είναι τι γίνεται όταν υπάρχουν συγκρούσεις μεταξύ θεμελιωδών δικαιωμάτων, δυνητικές συγκρούσεις ή πραγματικές συγκρούσεις μεταξύ των δικαιωμάτων που έρχονται από τη Χάρτα αφενός και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση αφετέρου, συγκρούσεις σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο αναφέρεται στο άρθρο 8, στο άρθρο 10, το δικαίωμα να υπάρχει μια αξιοπρέπεια και μια φήμη για κάθε πολίτη, το οποίο κατά κάποιο τρόπο έχει αποκομίσει μια ιδιαίτερη αυτονομία και συγκρούεται λιγάκι με το άρθρο 10 για την ε, ε, ελευθερία έκφρασης. Και αυτά προκύπτουν και από την περίφημη υπόθεση Βαν Χάνοβερ κατά της Γερμανίας. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τις συγκρούσεις ερμηνείας για δικαιώματα τα οποία είναι κοινά στην Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, νομίζω ότι η νομολογία του ΕΔΑΔ και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του Λουξεμβούργου θα πρέπει να προχωρήσουν σε μια εναρμόνιση μεταξύ τους. Νομίζω ότι αυτή είναι μια σωστή πορεία, γιατί και η συνδίκη τη Λισαβόνα επιβάλλει μια διαδικασία προσέγγιση. Κατά τα άλλα, το θέμα αυτό των δικαιωμάτων είναι τόσο ευρύ, τόσο δύσκολα, που δεν νομίζω ότι μπορώ να κάνω τίποτα άλλο παρά από μια γενική παρατήρηση. Τώρα, σε ό,τι αφορά την εφαρμογή των πρωτοκόλων, επανέρχομαι σε κάτι που διάβασα με μεγάλη προσοχή στην έκθεση του κ. Ζακέ. Τα πρωτόκολλα τα οποία είναι συναφή μετά την προσχώρηση της Ευρωπαϊκή Ένωση και περιλαμβάνουν δικαιώματα τα οποία τη χάνουν εγγύηση από τη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, αυτά είναι τα οποία θα πρέπει να τύχουν κύρωση και σε ό,τι αφορά τη μη διάκριση, το πρωτόκολλο 12 τη Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που αντιμετωπίζει μια πολύ σημαντική επιταγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τη μη διάκριση και είναι τμήμα τη πάγια νομολογία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει στην περίπτωση αυτή, εμφορούμενη και από το πνεύμα των κειμένων τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη νομολογία, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι το, άρθρο, το, πρωτόκολλο 12 θα προχωρήσει σε μια κύρωση γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση και σημαντικό για οποιαδήποτε δημοκρατική κοινωνία. Ευχαριστώ. Αναρωτιέμαι αν θα ήθελα να λάβει το λόγο σε αυτό το σημείο. Come Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομο να απαντήσω στα ερωτήματα που τέθηκαν και δεν έχουν απαντηθεί ακόμα. Καταρχάς από τον εισηγητή, τον ίδιο, σε ό,τι αφορά το, τη μορφή των διαπραγματεύσεων από πλευρά Συμβουλίου Ευρώπης. Ε, η Επιτροπή Υπουργών θα αποφασίσει από αυτού. Νομίζω ότι η απόφαση αυτή θα εμπνευστεί από αυτά που, ακούσαμε με πολλού σήμερα, δηλαδή από την επιθυμία οι διαπραγματεύσεις αυτές να διεξαχθούν όσο το δυνατόν ομαλότερα και γρηγορότερα και προς το σκοπό αυτό ε, μπορεί ενδεχομένως να, να διαμορφωθεί μία ανεπίσημη ομάδα εργασίας για τις διαπραγματεύσεις, η οποία θα αποτελείται, για παράδειγμα, από έναν αριθμό εκπροσώπων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μία σειρά εκπροσώπων που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και φυσικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι και αυτή προσκεκλημένη για να συμμετάσχει σε μια τέτοια ομάδα εργασίας. Αυτό θα διασφαλίσει επίσης και τις καλές επαφές με τις ε, χώρες μέλη. Και φυσικά θα υπογραμμίσει και όσα ακούσαμε και από τον εκπρόσωπο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης. Θα είναι και τα δύο σώματα εξαιρετικά σημαντικά σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Δεύτερη απάντηση που θα ήθελα να δώσω σε σχέση με το ερώτημα του κυρίου Νταφ για το ποια θα είναι τα μαθήματα τα οποία μπορούμε να εξαγάγουμε από την εμπειρία του Συμβουλίου της Ευρώπης σε ό,τι αφορά την επικύρωση του πρωτοκόλλου υπαριθμών 14. Θα ήθελα να τονίσω ότι το θέμα της ε, επικύρωσης του πρωτοκόλλου υπαριθμών 14 αποτελεί, αν θέλετε, μία μοναδική πολιτική εμπειρία. Και θα πρέπει να θυμόμαστε ότι μόνο μία χώρα συμμετείχε στην διαδικασία αυτή και να έχουμε επίσης υπόψη μας ότι η κυβέρνηση της χώρας αυτής ήταν υπέρ της ε, ε, έγκαιρης ε, επικύρωσης. Δεν μπορώ να εξαγάγω γενικότερα μαθήματα λοιπόν από την εμπειρία αυτή. Θα ήθελα να θεωρήσουμε μάλλον ως κάτι μοναδικό, ως ένα μοναδικό παράδειγμα. Νομίζω ότι οι πιο πολλές χώρες μέλη πλέον θα εμπνευστούν από το γεγονός ότι σήμερα έχουμε μία μοναδική ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε μία ε, περιοχή για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλη την Ήπειρο, όπου και η Ένωση και τα 27 κράτη-μέλη θα δεσμεύονται από τα ίδια πρότυπα σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα παρακολουθούνται από το ίδιο δικαστήριο. Αν ε, τα τηρήσουμε λοιπόν όλα στην προπτική αυτή, όλα θα πάνε καλά για μια διαδικασία ε, διαπραγματεύσεων, την οποία ελπίζω πραγματικά να είναι και γρήγορη και ομαλή. Ευχαριστούμε ο κύριος Νταφ. Ευχαριστώ ιδιαίτερα για την περιγραφή του προβλήματος του πρωτοκόλου 14. Είναι ενθαρρυντικό αν είναι η εξαίρεση. Το διαπραγμάτευση για λογαριασμό μας. Η Κομισιόν θα διαπραγματευτεί ή η υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Όχι κράτη-μέλη. Όχι κράτη-μέλη. Ο καθηγητής Κριστόφερσον αν θέλει να δευτερολογήσει. Ευχαριστώ πολύ. Έγινε ερώτηση κατά πόσον η προσχώρηση στο πρωτόκολλο 12 θα κάνει το πρωτόκολλο εφαρμόσιμο εκτελέσουμε σε κράτη-μέλη. Η απάντηση είναι όχι. Το πρωτόκολλο 12, στο βαθμό που είναι κοινή ευρωπαϊκή προδιαγραφή και όρος, ήδη είναι τμήμα του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Από αυτή την άποψη λοιπόν η αρχή των μη διακρίσεων ισχύει για την νομοθεσία της Ένωσης. Αλλά το πρωτόκολλο το ίδιο δεν είναι δεσμευτικό για το Ενωμένο Βασίλειο στις υποχρώσεις του έναντι των άλλων κρατών. Και το ίδιο ισχύει για οποιοδήποτε άλλη υποχρέωση που μπορεί να έχει ή να μην έχει κάποια χώρα σε σχέση με υποχρώσεις της Ένωσης. Και γι' αυτό η προοπτική της Ένωσης θα πρέπει να είναι όλα τα δικαιώματα με βάση τη σύμβαση να ισχύσει. Και από εκεί και πέρα τα κράτη θα έχουν τις δικές τους υποχρώσεις. Αν αυτή είναι η προσέγγιση της Ένωσης, τότε η προσχώρηση θα είναι διάτρετη. Αυτή είναι η πολιτική πραγματικότητα σήμερα. Και γι' αυτό το πρωτόκολλο είναι γραμμένο με τον τρόπο που είναι γραμμένο. Γιατί δεν υπήρχε σύνδεση ανάμεσα στι υποχρώσεις της και τι υποχρώσεις των κρατών μελών. Το πρωτόκολλο λοιπόν ουσιαστικά πάσχει πολιτικά ή νομικά πάσχει για πολιτικούς λόγους, όπω θέλετε, όπως θέλετε ε, πείτε Ο κ. Μπράνς επίσης ε, ρώτησε πώς ορίζουμε τα ε, αντιτιθέμενα δικαιώματα Ας αφήσουμε άλλους να ορίσουν. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα. Έχετε δυο διαδηλωτέ. Θα πρέπει να προστατεύετε ο ένας έναντι του άλλου, τους διαδηλωτέ. Θα πρέπει να βρούμε μια γραμμή ανάμεσα στους δύο διαδηλωτέ να μην δίνουν μάχες στους δρόμους. Δηλαδή το ίδιο δικαίωμα ο καθένα, αλλά τα δικαιώματα του ενό, το δικαίωμα του ενό αντίθεση με το δικαίωμα του άλλου. Θα πρέπει να ορίσουμε ποια είναι τα όρια στην ελευθερία έκφραση. Καλή ιδέα θεωρητικά, αλλά πολύ δύσκολο στην πράξη. Γι' αυτό έχουμε γενικού κανόνε, γενικά δικαιώματα, γενική νομοθεσία και τα δικαστήρια ορίζουν τα όρια. Φυσικά, ένα κοινοβούλιο μπορεί να πει τη γνώμη του για μια συγκεκριμένη κατάσταση, πάμε χάρη ελευθερία έκφραση. Και αυτό θα ληφθεί υπόψη μετά από το δικαστήριο. Αυτός είναι ο ρόλο ένα κοινοβουλίου. Ή οποιοδήποτε κοινοβολική ενός κοινοβουλίου ή οποιασδήποτε κοινοβουλευτική συνέλευση, εθνικά κοινοβούλια κλπ. Επίσης, από τη μεριά των εισηγητών έγινε μια ερώτηση. Η, η Ένωση είναι συγκρίσιμη με ένα κράτος αφενός. Από την άλλη μεριά όμω υπάρχει και διαφορά για τους συνεναγόμενους. Αν θέλουμε να πάρουμε το θέμα στα σοβαρά. Αν υπάρχουν μια προσφυγή κατά ενός κράτους και το κράτος θα πρέπει να είναι υπεύθυνο, το κράτος θα, μπορεί να θα πρέπει να μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του και με την νομοθεσία της Ένωσης. Και αν η Κομισιόν θέλει να πει κάτι, μπορεί να παρέμβει ως τρίτος. Αυτό γίνεται εξάλλου. Αν δεν είναι το κράτος υπεύθυνο και είναι η Ένωση υπεύθυνη, τότε η προσφυγή θα πρέπει να γίνει κατά της Ένωσης και θα πρέπει να υπάρξει ένα μηχανισμός πώ θα μεταφερθούν οι ευθύνε από ένα κράτος στην Ένωση αν κάποιος κάνει προσφυγή εναντίον ενός λάθο διαδίκου. Δεν είμαι πάντω υπέρ του να υπάρχουν επιπλέον νέοι κανόνε για να βολευτεί κατά κάποιο τρόπο η Ένωση η Ένωση θα πρέπει, αν μπει, να λειτουργεί με τους ίδιους κανόνες που ίσχυαν ως τώρα. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Ο κύριος Νταφ ρώτησε ε, ο χάρτης και η Ένωση, αν υπάρχει μια συμβατότητα και αν υπάρχει κίνδυνος με προσχώρηση στην ΕΣΔΑ, η Ένωση τι θέση θα έχει ως προς τα ε, δικαιώματα, ως προς τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η αρμονία μεταξύ της Ένωσης και των προδιαγραφών της Χάρτας και των προδιαγραφών της Σύμβασης είναι περισσότερο παρόμοιες παρά ανόμοιες. Σήμερα βλέπουμε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο συχνά να υιοθετεί υψηλότερε προδιαγραφές από ότι η Ευρωπαϊκή ή από ΕΣΔΑ. Αυτό το επιτρέπει η χάρτα και μπορεί να συνεχιστεί, αλλά μπορεί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να μην θέλει να πάει τόσο, να προχωρήσει τόσο πολύ αργότερα, δεν ξέρω. Το πιθανότερο είναι στο μέλλον να έχουν περισσότερη αρμονία παρά λιγότερη αρμονία. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Ο δόκτωρ Κράμερ που είναι υπάλληλο της Κομισιόν σε θέματα δικαιοσύνη και ανθρώπινα δικαιώματα. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να δώσω μια σύντομη απάντηση καταρχήν στο ερώτημα το οποίο ετέθη από τον κύριο Μπρόμς. Πώς δηλαδή θα επηρεαστεί η θέση των κρατών μελών αν η Ευρωπαϊκή Ένωση προσχωρήσει σε ένα πρωτόκολλο που δεν έχει κυρωθεί από το αντίστοιχο αυτό κράτος μέλος. Η απάντηση στο θέμα αυτό βρίσκεται στο άρθρο 2 του πρωτοκόλλου 8 στη Συνθήκη της Λισαβόνας, δηλαδή ότι η θέση του κράτους μέλους δεν θα πρέπει να τροποποιηθεί με κανένα τρόπο από την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πρωτόκολλο αυτό. Αυτό το οποίο μπορεί να είναι ένα πρόβλημα είναι το άρθρο 216 παράγραφος 2 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προβλέπει ότι οι διεθνείς συμφωνίες που συνάπτονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι δεσμευτικές για τους θεσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά την δική μα άποψη και το τόνισε και η Επίτροπο Ρέντιν σήμερα το πρωί, είναι πάρα πολύ σημαντικό η διαδικασία προσχώρησης η συμφωνία προσχώρησης να περιλαμβάνει και ένα κανόνα βάσει του οποίου οι υποχρεώσεις οι οποίες έλκονται από τις ουσιαστικές διατάξεις για τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες θα προκύπτουν μονάχα επί τη βάση πράξεων που ενεκρίθηκαν από τους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τον τρόπο αυτό υπάρχει ο μηχανισμός αποσύνδεσης ο οποίος πλήρως εξασφαλίζει και ξέρουμε ότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα για τα κράτη-μέλη που διασφαλίζει πλήρως την θέση των κρατών μελών. Να είμαστε λοιπόν σαφείς ότι η θέση των κρατών μελών όχι μόνο δεν θα αλλάξει σε ό,τι αφορά το διεθνές δημόσιο δίκαιο, κάτι το οποίο φυσικά δεν μπορεί να γίνει, αλλά δεν θα τροποποιηθεί ούτε και σε επίπεδο του ευρωπαϊκού δικαίου. Δεν θα υπάρξουν λοιπόν νέες υποχρεώσεις που θα προκύψουν για τα κράτη-μέλη και τα κράτη-μέλη θα είναι δεσμευμένα σε επίπεδο θεμελιωδών δικαιωμάτων από αυτό το οποίο σήμερα ισχύει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης από την χάρτα και τις βασικές αρχές του ευρωπαϊκού δικαίου, αλλά η πρόσβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύμβαση, κατά την άποψή μας, δεν θα προσθέσει το παραμικρό στις υποχρεώσεις των κρατών μελών στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και είναι πολύ σημαντικό να το έχουμε αυτό υπόψη μας, διότι από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η πλήρης αποσύνδεση και έχει εξασφαλιστεί, τότε πρόκειται για μια καθαρά πολιτική επιλογή όπου μπορεί να υπάρξει μεγάλη ελευθερία και να αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ελεύθερα σε ποια πρωτόκολλα θέλει να προσχωρήσει. Αλλά θα πρέπει να διακριθούν τα δύο αυτά σημεία, να, να ξεχωριστούν για τις ε, μεμονωμένες επιφυλάξεις των κρατών μελών και τα πρωτόκολλα τα οποία πρέπει να προσπογράψει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι ακόμα για το μηχανισμό συνεναγόμενης Ευρωπαϊκής Ένωσης που το έθεσε ένα αμφιβόλο κύριος Κριστόφεσεν. Πιστεύουμε ότι αυτό θα πρέπει να είναι ακρογωνιαίος λίθος της προσχώρησης να έχει αυτό το δικαίωμα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί όπως τόνισε ο κύριος Τίμερμαν σήμερα το πρωί σε ό,τι αφορά τα θέματα ουσιαστικού δικαίου δεν θα προκύψει τίποτα το ουσιαστικό το οποίο θα προσθεθεί. Η πραγματική προσθέμενη αξία είναι σε επίπεδο δικονομικού δικαίου και στο γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορεί να συμμετέχει ως διάδικος στις ε, δικαστικές διαδικασίες και στα σώματα της σύμβασης. Από αυτή την άποψη ο μηχανισμός συνεν... συνεναγόμενης Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σημαντικός γιατί σε περιπτώσεις που είναι σημαντικές στην ομολογία έχουν καταλογιστεί πράξεις των κρατών μελών που είναι εφαρμοστικές νομοθετημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ίδια τα κράτη-μέλη. Θεωρείται δηλαδή ότι το κάθε κράτος μέλος είναι απόλυτα υπόλογο για τις πράξεις του ακόμα και αν είναι απλές μεταγραφές ή εφαρμογές υποχρεώσεων που προκύπτουν από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο λοιπόν με τη διαδικασία συνεναγόμενης Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση να υποστηρίξει το συμβατό των νομικών της κανόνων με την, τους κανόνες της σύμβασης, αλλά επίσης και ενδεχομένω, αν θεωρήσει το ΕΔΑΔ ότι υπάρχει κάποια παραβίαση των κανόνων αυτών της σύμβασης, θα δεσμεύεται από την απόφαση του ΕΔΑΔ η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί σε αυτή την περίπτωση θα εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργία του συστήματος της Σύμβασης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων γιατί τότε θα πρέπει ο εναγόμενος να αντλήσει όλα τα απαραίτητα συμπεράσματα από την απόφαση του ΕΔΑΘ. Αυτό δεν είναι ένα προνόμιο το οποίο δίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι για τον ενάγοντα ένα προνόμιο γιατί ο ενάγων θα έχει ένα δεύτερο εναγόμενο, ο οποίος θα έχει αστική ευθύνη σε αυτήν την περίπτωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν προσπαθεί να προστατεύσει τον εαυτό της από αγωγές, αλλά αντίθετα να εξασφαλίσει ότι υπάρχει σωστή αντανάκλαση της εσωτερικής της ενομής τάξης σε όλη αυτή τη διαδικασία. Ευχαριστούμε. Ο, καθηγητής Ζαμπόλ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. για το ένα συνεναγόμενο. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα για να δείτε γιατί είναι αναγκαίο. Πάστε το κείμενο της κράτησης του ΕΤΑ. Σε συνταγματικά δικαστήρια Γερμανίας και Ρουμανίας λένε ότι τίθεται θέμα. Το τέξτ, si c'est le texte communautaire qui est... Στην περίπτωση αυτή, εδώ υπάρχει αντίθεση είτε με τα θεμελιώδη δικαιώματα, είτε πρόκειται για τη χρήση που κάνουν τα κράτη-μέλη στο περιθώριο αξιολόγηση που έχουν αυτή τη data protection. Ας πούμε ότι κάπω κάνει προσφυγή κατά της Γαλλίας ή της Ιταλίας στο δικαστήριο με βάση το κείμενο αυτό. Δεν έχουμε ερμηνεία ποιο είναι το πεδίο εφαρμογής για τα κράτη-μέλη και το θεωρώ αυτονόητο η Ένωση να είναι σύνδικος στην περίπτωση που θεωρηθεί ότι το πρόβλημα δημιουργείται από κείμενο της Ένωσης και όχι από κείμενο του κράτους μέλους. Κοντεφαντέρ, κοντεφέντεν, συνεναγόμενος, μπορούμε να, βρούμε, να ψάξουμε να βρούμε τον τρόπο, αλλά πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα επιμερισμού των αρμοδιοτήτων. Αυτό ήταν το παράδειγμα για το data retention. Τώρα, για το πρωτόκολλο και τις επιφλάκεις των κρατών μελών. Ο εισηγητής το είπε κατά επανάληψη. Αυτό θα ισχύσει για την Ένωση στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της και για τα κράτη-μέλη, όπως λέει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, in the field of EU law. Δεν έχει άμεση επίπτωση στις εσωτερικές αρμοδιότητες των κρατών μελών. Έχει επίπτωση μόνο στο πεδίο εφαρμογής του κοινωτικού δικαίου. Η Ένωση μπορεί να επιλέξει ό,τι θέλει ανησύχησα λίγο για αυτά που είπε το πρωί. Με πολύ σαγίνη η κυρία Ρέντιν για τις δύο φάσεις. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ πώς ε, προσχωρώντας κανείς στην ΕΣΔΑ δεν, δεν προσχωρεί και στο πρωτόκολλο. Μου είναι αδιανόητο αυτό. Αν η Κομισιόν μας λέει τώρα ότι στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων θα μελετήσουμε και τα πρωτόκολλα, χρήσιμο. Αλλά αν είναι μετά στις ελληνικές καλέμβες δημιουργεί σοβαρό πρόβλημα. Διότι υπάρχουν στοιχεία εκ των όνου κάνευ και τα έχει χρησιμοποιήσει ήδη τα στοιχεία αυτά το δικαστήριο, αλλά ήδη μακρηγόρησε. Πρόεδρος, ευχαριστούμε και τελειώσαμε με αυτή την πρώτη φάση της συνάντησης και τώρα ερχόμαστε στη δεύτερη και τελευταία φάση και αρχίζουμε με τον καθηγητή Francis Jacobs, καθηγητή στο Λονδίνο, King's College και γενικό εγγελέα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και χαίρομαι που έχω την ευκαιρία να έρθω εδώ στην Επιτροπή σας σήμερα για να προσπαθήσω να απαντήσω κάποια από τα πολύ ενδιαφέροντα ερωτήματα. Σημείο κίνησης μου θα είναι η, η πρόταση ψηφίσματος και νομίζω ότι χρήσιμο θα είναι να κοιτάξουμε τα θέματα με τη σειρά που εμφανίζονται στο ψήφισμα. Αλλά και φυσικά να λάβουμε υπόψη κάποιες από τις ιδέες οι οποίες ε, ακούστηκαν σήμερα, κάποια από τα επιχειρήματα τα οποία προβλήθηκαν. Εν συντομία, τα επιχειρήματα υπέρ της προσχώρησης που αναφέρονται στην παραγράφη 1 όπως τονίστηκε ήδη, τώρα που υπάρχει υποχρέωση προσχώρηση στη σύμβαση, δεν χρειάζεται να προσπαθήσουμε να πείσουμε υπέρ της προσχώρησης. Άρα τα επιχειρήματα υπέρ της προσχώρησης έχουν σημασία τώρα γιατί μπορεί να θέσουν τους όρους, αν θέλετε, που θα επηρεάσουν την προσχώρηση και ενδεχόμενους περιορισμούς σε ό,τι αφορά την προσχώρηση, πέρα από τα συμβολικά επιχειρήματα τα οποία αναφέρονται στην πρώτη υποπαράγραφο και να επικεντρωθούμε πραγματικά στην ανάγκη προσχώρησης με αποτελεσματικό τρόπο για να δοθεί προστασία σε ό,τι αφορά τα μέτρα που λαμβάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχω την εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει, και αυτό θα πρέπει να αποτελεί και ο στόχο, το στόχο της ε, διαδικασίας να βρίσκεται το δυνατόν όσο πιο πολύ γίνεται στην ίδια κατάσταση, στην ίδια θέση με τα κράτη-μέλη. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν ε, γενικές εξαιρέσεις, γενικές επιφυλάξεις σε ό,τι αφορά τον ε, έλεγχο, να υπάρχουν μόνο ό,τι είναι απολύτω απαραίτητο υπό το φως των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την κατανομή ε, αρμοδιοτήτων μεταξύ Ένωσης και κρατών μελών. Θα επανέλθω στο θέμα αυτό. Όπως ξέρουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ήδη υποκείμενο δικαίου και δεσμεύεται για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε ό,τι αφορά και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, παρά το γεγονός ότι δεν είναι ακόμα μέλος η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά βασικός ε, στόχος της προσχώρησης, έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει να είναι να δοθεί αν θέλετε, με το σύστημα της σύμβασης μια, ένα δικαστικό ένομο μέσο. Αυτό θα είναι η προστιθέμενη αξία και αυτό ισχύει ιδιαίτερα υπό το πλαίσιο της συνθήκης της Λισαβόνας γιατί το δικαστήριο δεν έχει δικαιοδοσία για να αποφανθεί. Όπως ξέρετε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ε, δεν μπορεί να αποτελέσει νομικό μέσο σε ορισμένες περιπτώσεις, είτε πρόκειται για πρωτογενές δίκαιο, για παράδειγμα, όπου το ε, δικαστήριο δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά του, είτε επειδή, επειδή ένα άτομο δεν έχει το απαραίτητο κύρος για να προς, ε, προσάγει μια υπόθεση στο δικαστήριο. Αλλά έχω την εντύπωση ότι το δικαστήριο στο Στρασβούργο θα πρέπει να ασκεί δικαιοδοσία σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, πρωτογενές δίκαιο. Δεν θα πρέπει να, να εξαιρεθεί αυτό από τη δικαιοδοσία του δικαστηρίου του Στρασβούργου. Θα πρέπει να αποτελεί ένα από τα ωφέλη, αν θέλετε, της διαδικασίας αυτής. Και είναι δυνατόν αυτό να ενθαρρύνει το ΔΕΚ να επεκτείνει τη δική του δικαιοδοσία. Γιατί φυσικά είναι πιο χρήσιμο να γίνεται τέτοια εκδίκαση από το ΔΕΚ σε πρώτη φάση, σε πρωτοβάθμιο επίπεδο, πριν φτάσουμε στο δικαστήριο του Στρασβούργου. Και δεν έχω την εντύπωση ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα στον επιτραπή στο ΕΔΑΔ να ε, αποφαίνεται για πρωτογενές δίκαιο, γιατί σε κάποιες περιπτώσεις υπονοήθηκε ότι αυτό ενδεχομένως να έδινε στο ΕΔΑΔ τη δυνατότητα να ακυρώσει το πρωτογενές δίκαιο της Ένωσης. Αυτό προφανώς δεν ισχύει. Δίδοντας ε, τέτοια δικαιοδοσία στο ΕΔΑΔ, δεν θα επιτρέψει στο δικαστήριο αυτό να ακυρώσει τέτοιες πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν πρόκειται να ακυρωθούν τέτοιες ε, πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπινών Δικαιωμάτων. Εγώ θεωρώ, αντίθετα με αυτά που είπαν άλλοι, ότι το δικαστήριο του ΕΔΑΔ δεν θα μπορεί καν να αποφανθεί επί της συμβατότητας ε, με τη σύμβαση. Απλά θα αποφασίσει κατά πόσο δεν θα συμπεριληφθεί δηλαδή κάποια γενική απόφαση, δικαστική απόφαση για τα γεγονότα. Αυτό είναι μια αρμοδιότητα της ίδιας της Ένωσης, το πώς αντιδράσει δηλαδή στη δικαστική απόφαση. Ούτε πρόκειται να προκληθεί ανάκληση των μέτρων, γιατί τα μέτρα θα μπορούσαν να εφαρμοστούν και να ερμηνευτούν με διαφορετικό τρόπο. Άρα δεν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα στο να δοθούν τέτοιες ευρύτερες αρμοδιότητες στο ΕΔΑΒ σε ό,τι αφορά το θέμα των ορμοδιοτήτων, το οποίο εξετάζεται στην επόμενη παράγραφο του ψηφίσματος, τα πράγματα είναι παρόμοια. Καταρχάς, θα ήθελα να πω ότι η προσχώρηση δεν θεωρώ ότι περιλαμβάνει διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της Ένωσης και δεν δημιουργεί γενικότερη αρμοδιότητα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό φαίνεται ότι δυστυχώς αποτελεί μια ευρεία παρανόηση. Είναι σαφέ από την ίδια τη συνθήκη ότι δεν υπάρχει τέτοια διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω προσχώρηση. Και όπως είπε και ο καθηγητής ε, Ζακή, δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ του κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται να σεβαστεί ε, μεμονωμένα δικαιώματα και κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αρμόδια για τέτοια δικαιώματα. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά το δικαίωμα της ανεξιθρησκείας. Αυτό είναι κάτι το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη δεσμεύεται να σεβαστεί. Και υπήρχαν περιπτώσεις όπου το δικαστήριο έχει αποφανθεί ότι υπάρχει δικαίωμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση να σεβαστεί το δικαίωμα αυτό. Δεν σημαίνει αυτό όμως ότι υπάρχει νομοθετική αρμοδιότητα της Ένωσης επ' αυτού. Αυτό, αυτό αποτελεί απλά μία παρανόηση. Η αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να αποφασίσει για την προσχώρηση. Στο μέλλον η Ένωση θα πρέπει να πληρεί του όρου που έχουν αποφασιστεί από το δικαστήριο για τη συνθήκη. Θα περιοριστούν δηλαδή οι αρμοδιότητέ τη. άρα ούτε εκεί υπάρχει πρόβλημα λόγω τη προσχώρηση στην σύμβαση. Νομίζω ότι το ίδιο ισχύουν λίγο πολύ και σε ό,τι αφορά τα πρωτόκολλα. Και πάλι έχω την εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να συμμορφωθεί με τι ε, απαιτήσει περί συμμόρφωσης της Ένωσης ε, με, το, με τη Σύμβαση, θα πρέπει να φέρει όλα τα κράτη-μέλη και να τα κάνει μέρη του πρωτοκόλλου όσο γίνεται. Και πάλι υπό τον όρο ότι το γεγονός ότι η Ένωση γίνεται μέρος των πρωτοκόλλων και ότι δεν υποβάλλει ενστάσεις και επιφυλάξεις δεν σχετίζεται με τα κράτη-μέλη τα οποία δεν είναι μέλη του πρωτοκόλου, των πρωτοκόλων ή έχουν εκφράσει επιφυλάξεις στα πλαίσια των πρωτοκόλων. Μπορεί κάποια τα δικαιώματα να μην σχετίζονται απαραίτητα με το έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για παράδειγμα το δικαίωμα στη ζωή, το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν φανταζόμαστε, δεν είναι πιθανό να παραβιάσει. Αυτό και επίσης δεν υπάρχει λόγος η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην προσχωρήσει στα πρωτόκολλα. Σε ό,τι αφορά δηλαδή πρωτόκολλα που δεν σχετίζονται άμεσα με το έργο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εγώ δεν θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποφύγει την υποχρέωση δέσμευσης στην παρούσα φάση σε ό,τι αφορά την προσχώρηση στα πρωτόκολλα και να έχει ένα γενικό δικαίωμα προσχώρηση σε μετέπειτα φάση, γιατί μόνο η παρανόηση αυτή του ποιο θα είναι, ποιος θα είναι ο αντίκτυπος της προσχώρησης στα πρωτόκολλα επικρατεί. Και καλό θα ήταν ο κόσμος να καταλάβει τι σημαίνει η επικύρωση των πρωτοκόλων και ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε ένσταση για την επικύρωσή τους. Ε, Επιπρακτικών ζητημάτων τώρα ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων και σε ό,τι αφορά την Επιτροπή Υπουργών σε ό,τι αφορά την παράγραφη παριθμών 5 του ψηφίσματος. Η τοποθέτηση αυτή μου φαίνεται αρκετά άμεση. Φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει δικαίωμα να υποβάλει υποψήφιους δικαστές, γιατί ε, σε πολλές περιπτώσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι διάδικος ενώπιον του δικαστηρίου και εν μέρη επειδή θα είναι εκπρόσωπος ε, του νομικού συμβουλίου του Συμβουλίου της Ευρώπης. Επίσης δεν υπάρχει λόγος γιατί δεν υπάρχει λόγος να περιοριστεί ο ρόλος των δικαστών. Θα πρέπει να ισχύει το συνηθισμένο σύστημα της ε, σύμβαση. Κατά τρίτον, πώς θα πρέπει να ορίζονται οι δικαστέ από πλευρά τη Ένωση και πάλι ακολουθώντα στο βαθμό του δυνατού το φυσιολογικό σύστημα άσχετα από τις ε, θεσμικές ε, ρυθμίσεις οι τρει υποψήφοι θα ορίζονται με κάποια διαδικασία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να, ακολουθούν, να και να τηρούνται οι απαραίτητες ε, δικλείδες ασφαλείας, να υπάρχει η απαραίτητη διαφάνεια για τις υποψηφιότητες αυτές και πρέπει να ομολογήσω ότι προσωπικά δεν θεωρώ ότι υπάρχει ανάγκη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διορίζει μέλη στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ε, υποβολή υποψηφιότητα των δικαστών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να συμμετάσχει σε άλλους, με άλλους τρόπους στη διαδικασία αυτή. Μια νέα διαδικασία της συνθήκης της Λισαβόνας yeah. τους δικαστές και τους εισαγγελείς. Είναι σημαντικό λοιπόν να υπάρχει η παρουσία υποψηφίων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη διαδικασία επιλογής τους μπορούν να παίξουν κάποιο σημαντικό ρόλο και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία επιλογής των δικαστών μέσα στην Ανεξάρτητη Επιτροπή. Τέλος, σε ό,τι αφορά την Υπουργική Επιτροπή, νομίζω ότι είναι πρόδειλο ότι θα πρέπει να εκπροσωπείται και στην Υπουργική Επιτροπή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενδεχομένως θα πρέπει να εκπροσωπείται σε όλες τις περιπτώσεις που έχει να συνεδριάσει η Επιτροπή Υπουργών, όχι μονάχα στην λήψη αποφάσεων, αλλά και στη διαδικασία εκτέλεσης των αποφάσεων. Γι' αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να την χάνει εκπροσώψεις από την πλευρά της Κομισιόν, μέσω της Κομισιόν. Το θέμα των προσφυγών μεταξύ κρατών που αναφέρεται στην παράγραφο 6 είναι ένα ακαθόδες θέμα. Ίσως ένα από τα πιο δύσκολα θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Φαίνεται ότι θα ήταν ορθό, χωρίς να σας εξηγήσω ακριβώς γιατί, να αποκλείσουμε τις προσφυγές μεταξύ κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά θέματα ευρωπαϊκού δικαίου, σε σχέση με θέματα τα οποία μπορεί να εμπλέκουν μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά υπάρχουν κάποιες δυσκολίες που μπορώ να δω εδώ. Πρώτα απ' όλα δεν είναι σαφές για μένα ότι η τωρινή συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το άρθρο 344, ότι αποκλείει απόλυτα αυτές τις διακρατικού χαρακτήρα προσφυγίας. Έχει αναφερθεί το άρθρο 34, λέει τα κράτη-μέλη δεσμεύονται να μην υποβάλουν ε, προσφυγές σε σχέση με την εφαρμογή ή την ερμηνεία των συνθήκων σε οποιοδήποτε άλλο φορέα, εκτός από αυτό που προβλέπεται από τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι η διαδικασία στο ΕΔΑΤ δεν είναι μία από αυτές που προβλέπονται μέσα από την συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή που θα προσχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην ΕΣΔΑ, στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Δεύτερο πρόβλημα, ότι αν υπάρξει προσπάθεια να υπάρξει αποκλεισμό μόνο στις περιοχές που εμπλέκεται η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό ήταν ένα πολύ δύσκολο κριτήριο στην εφαρμογή του και ποιος θα αποφάσιζε πώς θα εφαρμοζόταν. Και πάλι θα μπορούσε κανείς να διαφυσβητήσει την εφαρμογή του από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων γιατί αυτό θα δημιουργήσει πρόβλημα κατανομής αρμοδιοτήτων. Είναι δύσκολο θέμα, αλλά εγώ πρέπει να σας ομολογήσω ότι για μένα είναι ένα γενικό θέμα. Δεν θέλουμε τώρα να αντιμετωπίσουμε όλες τις δυνητικές δυσκολίες οι οποίες μπορούν να προκύψουν. Υπάρχει μια τάση, υπάρχει ένας κίνδυνος να βλέπουμε παντού δυσκολίες και να προσπαθούμε να τις ρυθμίσουμε από τώρα. Ενώ μια καλύτερη λύση είναι να αφήσουμε αυτά τα προβλήματα και να τα αφήσουμε στην πράξη να επιληθούν. Αν δει κανεί πώ θα λειτουργήσει το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Λουξεμβούργου ή και το ΕΔΑΘ να λύσουν προβλήματα που δεν προσβλεπόταν στην ΕΣΔΑΔ ή στη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης <clears throat> με ικανοποιητικό τρόπο, τότε όλα αυτά θα πρέπει να μας γεμίσουν και σε, με μια μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην πρακτική των δικαστικών και στην πρακτική των κρατών μερών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν προσπαθούν να επιλύσουν όλα αυτά τα δύσκολα θέματα ήδη εκ των προτέρων. Κάτι ακόμα όμως το οποίο νομίζω για μένα ότι είναι σαφές είναι ότι όταν υπάρχει μια προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που εμπλέκει την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα ήταν επιθυμητό, θα ήταν ίσως απαραίτητο το εμπλεκόμενο κράτος μέλος ή και τα εμπλεκόμενα κράτη-μέλη, καθώς και η Ευρωπαϊκή Ένωση η ίδια, να είναι συνεναγόμενη, να είναι συνδιάδικη μάλλον, στη διαδικασία ενώπιον του ΕΔΑΔ. Μπορεί να μην είναι εξ αρχής σαφές ποια θα πρέπει να είναι η σωστή διάκριση αρμοδιοτήτων μεταξύ ΕΔΑΔ και Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, μόνο στο τέλος μιας διαδικασία μπορεί να διαφανεί αυτό σαφέστερα. Αλλά για μένα αυτό δεν αποτελεί ένα πρόβλημα, γιατί το ΕΔΑΔ φυσιολογικά δεν θα χρειαστεί να κάνει μία διάκριση αρμοδιοτήτων. Η δική του αρμοδιότητα είναι να, κατα... να αποφασίσει αν υπήρξε μια παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά δεν είναι υποχρεωμένο να αποφασίσει ποιο είναι ο φορέα ο οποίο είναι υπεύθυνο για αυτή την παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η περίπτωση Μπόσφορου ήταν σαφή σε αυτή την περίπτωση. Θα μπορούσε να αποφασίσει ότι υπήρξε μια παραβίαση, αλλά θα μπορούσε να αφήσει μετά στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αποφασίσει πού θα έπρεπε, με ποιο τρόπο θα έπρεπε να αποδοθεί η κατάλληλη θεραπεία προς τον ενάγοντα. Επομένως λοιπόν δεν θεωρώ ότι αυτό είναι ένα ανυπέρβητο πρόβλημα. Νομίζω ότι ξεπέρασε και το χρόνο μου. Έχω ξεπεράσει το χρόνο μου λοιπόν. Έχω μερικές λεπτομέρειες ακόμα να προσθέσω και συγγνώμη για την καθυστέρηση. Κλείνοντας, θέλω να κάνω δύο γενικές παρατηρήσεις. Μου φαίνεται καταρχήν ότι σε αυτή τη διαδικασία προσχώρησης θα πρέπει να προσπαθήσουμε να έχουμε τις λιγότερες δυνατές τροποποιήσεις στα, στις συμβάσεις και τη συνθήκη. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε πρόσθετες δυσκολίες, δεν θέλουμε να αλλάξουμε τα πράγματα εάν δεν είναι απαραίτητο. Προσωπικά λοιπόν, εγώ δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ειδική θεραπεία, ένα ειδικό σύστημα προσφυγής ενώπιον του ΕΔΑΔ, ώστε να μπορεί το ΕΔΑΔ να έχει τον πρώτο λόγο. Έτσι και εδώ δεν νομίζω ότι συμβαίνει αυτό, γιατί υπάρχουν πράξεις πρωτογενούς δικαίου που δεν μπορούν να εξεταστούν από το ΕΔΑΔ. Υπάρχουν περιοχές που δεν έχει αρμοδιότητα και δοσηδικία το ΕΔΑΔ. Ακόμα και εκεί που έχει τέτοια δοσηδικία δεν υπάρχει κάποια υποχρέωση να παραπέμπεται αυτό το θέμα να παραπέμπεται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, παραδείγματο χάρη, ένα θέμα που του φτάσει στο ΕΔΑΔ. Και το τελευταίο σχόλιο που θέλω να κάνω, το τελευταίο και, τελευταίο και σημαντικό όμως που είναι ίσως αφιλεγόμενο, μου φαίνεται ότι η ΕΣΔΑ, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, θα πρέπει να θεωρηθεί το κύριο πρότυπο ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ακόμα και μετά την εφαρμογή και την συμπερίληψη τη συνθήκη τη Λισαβόνα τη Χάρτα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Μπορεί να είναι ευρύτερη η χάρτα, μεν, αλλά τα δικαιώματα τη χάρτα που αντανακλούν αυτά τα οποία αποφάσει η συνέλευση που αντανακτούν αυτά τη σύμβαση δεν ερμηνεύονται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο όπως η σύμβαση. Α θυμόμαστε επίση ότι η εμβέλεια τη χάρτα είναι ακόμα πολύ περιορισμένη. Αναφέρεται μόνο στα θεσμικά όργανα και τα σώματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μόνο όταν εφαρμόσουν κοινοτικό δίκαιο. Και δεν είναι εύκολο πάντα αυτό κανεί να το διακριβώσει αν ισχύει ή όχι. Και φυσικά η χάρτα δεν έχει καμία εφαρμογή στα 20 κράτη του Συμβουλίου της Ευρώπης που δεν είναι μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά έχουν υπογράψει την Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Για να μην υπάρξει λοιπόν κατακαιρματισμό των προτύπων ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρώπη, πιστεύω ότι θα ήταν επιθεμητό να θεωρήσουμε ότι η Σύμβαση η ΕΣΔΑ είναι το κυριότερο εργαλείο και επομένως είναι σημαντικό η προσχώρηση της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ΕΣΔΑ να ενισχύσει και όχι να αποδυναμώσει αυτή τη σύμβαση. Σας ευχαριστώ. τελευταία παρέμβαση τη κυρία Άννας Μπενάκη, που υπήρξε πρόεδρο του ε, Ελληνικού Κοινοβουλίου και καθηγητής τη Νομική Σχολή Κοινωνικών Αθηνών. Έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε το λόγο και θέλω να τον χρησιμοποιήσω στην αρχή για να συγχαρώ θερμά τους οργανωτές αυτής της ε, ακρόασης και για τον τρόπο που την οργάνωσαν. Είμαι βέβαια η τελευταία στη σημερινή ακρόαση και έχω είτε το ευμενές είτε το δυσμενές προνόμιο να έχουν λεχθεί σχεδόν όλα όσα ε, ανήκουν στο θέμα αυτό τόσο πολύ που ό,τι θα πω σε λίγο να μοιάζει σαν να πρόκειται να κομίσω γλάφκα εις Αθήνας. Ε, η προετοιμαζόμενη πάντως προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου είναι όπως έχει επισημανθεί ένα γεγονός με μεγάλη συμβολική, πολιτική και θεσμική σημασία. Ο συμβολισμός και η θετική πολιτική διάσταση του εγχειρήματος έχουν επισημανθεί από πολλές πλευρές Στη φάση όμως αυτή μας απασχολεί πιο συγκεκριμένα η θεσμική διάσταση της προσχώρησης, καθώς η προσχώρηση αυτή συνεπάγεται πρώτα απ' όλα την ανάγκη εναρμόνισης του τρόπου με τον οποίο οι δύο ευρωπαϊκές ένομες τάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ε, Συνθήκης της ΕΣΔΑ, τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι δύο προσεγγίζουν, ερμηνεύουν και εφαρμόζουν το υπάρχον δίκαιο προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Αυτή είναι μια αναγκαία εναρμόνιση στο ουσιαστικό δίκαιο. Όμως αναγκαία είναι η εναρμόνιση και στις ακολουθούμενες διαδικασίες επιδίωξης και επίτευξης της προστασίας των δικαιωμάτων του πολίτη, τις οποίες εφαρμόζουν οι δύο πλευρές, ανάλογα με το δικονομικό σύστημα της κάθε μιας. Αυτή είναι η αναγκαία εναρμόνιση στο δικονομικό δίκαιο. Και τέλος υπάρχει ανάγκη προσαρμογής στη σύνθεση και στον τρόπο λειτουργίας ορισμένων θεσμικών οργάνων της ΕΣΔΑ ε, κατά το μέτρο που έχουν ως αντικείμενο την προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ασχολούμε πρώτα με την εναρμόνιση στο ουσιαστικό δίκαιο, τονίζοντας ότι ο χάρτης θεμελιωδών ε, δικαιωμάτων που ενσωματώθηκε από άποψη ισχύω στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση απομάκρυνε σημαντικά τον κίνδυνο επικαλύψεων, παρερμηνεών και συγκρούσεων. Το άρθρο 51 παράγραφος 1 του χάρτη και το 52 παράγραφος 3 με το γνωστό τους περιεχόμενο εξουδετερώνουν τις περισσότερες πιθανές αιστείες σύγκρουσης. Οι διατάξεις αυτές συμπληρώνονται από το προήμιο και τις επεξηγήσεις του χάρτη, οι οποίες παραπέμπουν για την ανέβρεση της ακριβούς ενίας του δικαιώματος στην ε, νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του Στρασβούργου και ε, στην νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, η εξομάλυση αυτή στο ουσιαστικό πεδίο έχει βρει πράγματι την αντιστοιχία της και στην ομολογία των δύο ευρωπαϊκών δικαστηρίων. Η εξέλιξη της ομολογίας τους και η φυστάμενη μεταξύ των δικαστηρίων αυτών συνεργασία ε, δίνουν πολλές ελπίδες για την επίτευξη κατά το δυνατόν πλήρους εναρμόνισης. Πρώτα απ' όλα η νομολογία του Δικαστηρίου του Λουξεμβούργου από τη μία πλευρά εμφανίζει μια σταθερή τάση να ακολουθεί σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων την ΕΣΔΑ, σχεδόν σαν να ήταν ισχύον δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και να προσφεύγει στη σχετική νομολογία του Δικαστηρίου του Στρασβούργου. Ως πλέον χαρακτηριστική αξίζει να αναφερθεί η γνωστή απόφαση Ισπανίας κατά Ηνωμένου Βασιλείου του 2006, όπου το Δικαστήριο του Λουξεμβούργου αντιμετωπίζοντας προσφυγή της Ισπανίας κατά του Ηνωμένου Βασιλείου επί θέματος ε, τον αποκλεισμό του Γιβραλτάρ από τις ευρωπαϊκές εκλογές, το οποίο είχε κριθεί από το δικαστήριο του Στρασβούργου με την απόφαση Μάθιους εναντίον ε, Ηνωμένου Βασιλείου του 1999 ως συμπεριφορά αντίθετη με την ΕΣΔΑ. Απέρριψε λοιπόν το, το δικαστήριο του Λουξεμβούργου την ε, προσφυγή ε, της ε, Ισπανίας με την αιτιολογία ότι έπρεπε να εφαρμοστεί η απόφαση Μάθιους του Δικαστηρίου του Στρασβούργου. Εδώ βέβαια τίθεται ένα ερώτημα εάν παίρνει και θέση στον έλεγχο του πρωτογενούς δικαίου από το Δικαστήριο του, ε, του Στρασβούργου. Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι όμως από την άλλη πλευρά η νομολογία του Δικαστηρίου του Στρασβούργου σε σχέση με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την νομολογία του Δικαστηρίου του Λεξεμβούργου. Και πάλι ενδεικτικά και μόνο αξίζει να αναφερθεί η γνωστή απόφαση Ζολοτούκιν versus εναντίον Ρωσίας του 2009 όπου το Δικαστήριο του Στρασβούργου προκειμένου να καθορίσει την έννοια του κανόνα «ne bis in idem» και ιδίως την έννοια του «idem», κανόνα ο οποίος ισχύει και στο πλαίσιο του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως παραδείγματος χάρη στο δίκαιο του ανταγωνισμού ή στο δίκαιο της συνθήκης Schengen, Κατέληξε λοιπόν να δεχθεί την έννοια που επεκράτησε στο πλαίσιο του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι δηλαδή απαιτείται ταυτότητα των πραγματικών γεγονότων. Και έτσι έδωσε και τέρμα στη μέχρι τότε εκφερόμενη και μάλλον αμφιταλαντευόμενη νομολογία του. Και πολύ πιο σημαντική είναι η γνωστή ε, απόφαση ε, Μπόσφορους εναντίον Ιρλανδίας του 2005, η οποία δέχθηκε την ύπαρξη τεκμηρίου ισοδύναμης προστασίας των ανθρωπίνων ε, δικαιωμάτων από το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το δίκαιο της ΕΣΔΑ. Πλην όμως το τεκμήριο αυτό είναι μαχητό όπως είπε και ανατρέπεται όταν η προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπό τις συγκεκριμένες περιστάσεις της κρινόμενης περίπτωσης αποδεικνύεται ως εμφανώς ανεπαρκής. Βέβαια στο σημείο αυτό αρχίζει μια καινούργια συζήτηση για το πότε και πώς κρίνεται το εμφανώς ανεπαρκής, την οποία δεν μπορούμε να εισέλθουμε τώρα. Φυσικά παραμένουν ακόμη αποκλίσεις των δύο ενόμων τάξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ΕΣΔΑ στο ουσιαστικό δίκαιο. Όπως παραδείγματο χάρη στο προνόμιο της ε, μη ενοχοποίησης, ε, το οποίο εφαρμόζεται σε ευρύτερη βάση από το Δικαστήριο του Στρασβούργου βάσει του άρθρου 6 της ΕΣΔΑ. Σύμφωνα με την ομολογία αυτή, το ε, προνόμιο καλύπτει πάσης φύσεως δηλώσεις, έστω και έμεσες πληροφορίες, ε, ευρύτερα από ότι στο δίκαιο του ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που περιορίζεται μόνο σε δηλώσεις ευθέως ενοχοποιητικές όπως επίσης υπάρχουν αποκλήσεις στην εφαρμογή των ε, διατάξεων περί ασύλου ως προς την προσωρινή κράτηση είναι ενδιαφέρον το δικαστήριο του Στρασβούργου δέχθηκε νόμιμη την επταήμερη κράτηση του ετούντος άσυλο, ενώ στο δίκαιο αντιθέτως της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, απαγορεύεται κάθε κράτηση ή και στο δίκαιο της απέλασης ε, και ιδιαίτερα του κριτηρίου που χρησιμοποιείται για την απέλαση ε, και στην ΕΔΑ ε, κρατούνται, υπάρχουν διαφορές ως προς το ποιο είναι το κριτήριο που χρησιμοποιείται για να θεωρηθεί απαγορευμένη η απέλαση. Εάν θα δοθεί έμφαση στην υπηκότητα όπως συμβαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή εάν θα δοθεί έμφαση όπως συμβαίνει με την ΕΣΔΑ, με το Δικαστήριο του Στρασβούργου, εάν ε, το κριτήριο αυτό δεν είναι η υπηκότητα αλλά είναι ο βαθμός ένταξης του ε, στο φιλοξενούν κράτος. Εν πάση περιπτώσει, γεγονός είναι ότι η νομοθετική και νομολογιακή εναρμόνιση στο πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των δύο ενόμων τάξεων και της αντίστοιχης νομολογίας των δικαστηρίων είναι τόσο προχωρημένη ε, ώστε να πρέπει η ανάλογη πρόοδος να επιτευχθεί και στα λοιπά ερωτήματα που θέτει η ενδεχόμενη προσχώρηση, δηλαδή στη διαδικαστική εναρμόνιση, ιδίω σε σχέση με τα δύο ευρωπαϊκά δικαστήρια και τη διαμόρφωση των θεσμικών οργάνων της ΕΣΔΑ. Πιστεύω μάλιστα ότι αν η εναρμόνιση στο ουσιαστικό δίκαιο φτάσει σε ένα ιδεώδες σημείο, τα άλλα θέματα που ανέφερα λύνονται περίπου αυτομάτως. Εν πάση περιπτώσει ως προς την κατάστρωση και εναρμόνιση των διαδικασιών ε, ενώπιον του Δικαστηρίου του Στρασβούργου ανακύπτουν ορισμένα ερωτήματα ε, ως προς το αντικείμενο της δίκης ενώπιον του Δικαστηρίου του Στρασβούργου, ως προς τους συμμετέχοντες στο δικαστήριο αυτό, τους διαδίκους και ως προς τη σχέση μεταξύ των δύο Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων. Πρώτα, ως προς το αντικείμενο της δίκης, είναι σαφές ότι το Δικαστήριο του Στρασβούργου ερευνά από αφορμή ατομική προσφυγή την πιθανή παραβίαση της ΕΣΔΑ πρώτον εκ μέρους κράτου, κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης ε, δεύτερον από πράξεις, ε, την παραβίαση από πράξεις των οργάνων της Ένωσης, πάσης φύσεως μέτρα ή διοικητικέ και νομοθετικές πράξεις του δευτερογενούς δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το τρίτο που ερωτάτε είναι ελέγχεται από το δικαστήριο του Στρασβούργου και η συμφωνία ή μη συμφωνία του πρωτογενούς δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως αυτό τυποποιείται στη συνθήκη με την Ευρωπαϊκή Ένωση της συμφωνίας με την ΕΣΔΑ. Η τελευταία περίπτωση αυτή είναι προβληματική για πολλούς λόγους, όπως διότι θέτει μεταξύ άλλων και το θέμα δικαιοδοσίας μεταξύ των δύο δικαστηρίων, καθώς επίσης διότι ανοίγει και το ενδεχόμενο εισχώρησης της, της αρμοδιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πράγμα που αντιβαίνει στη συνθήκη και στο άρθρο 6 παράγραφος 2 και παρακολούθησα με πολύ ενδιαφέρον τις θέσεις του καθηγητού κυρίου Τζέικοψ που τώρα υπήρξε πολύ σαφής ε, και πρότεινε την υπαγωγή και του πρωτογενούς δικαίου της Ένωσης στην αρμοδιότητα του Δικαστηρίου του Στρασβούργου. Και όταν λέμε του πρωτογενούς δικαίου εννοούμε μόνο τις διατάξεις της συνθήκης αυτής καθεαυτής και τις νομοθετικές πράξεις που έχουν όμως ισοδύναμη ε, δύναμη με τις ε, διατάξεις της συνθήκης. Ενώ έξω μένουν και είναι δευτερογενές δίκαιο η κοινή νομοθετική παραγωγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες αποφάσεις. Λοιπόν, το ερώτημα είναι τι θα γίνει με το πρωτογενές δίκαιο με την περιορισμένη έννοια που το έθεσα. Μου φαίνεται ότι η ενδεδειγμένη λύση θα ήταν το δικαστήριο του Στρασβούργου να απέχει από την κρίση αυτή και να την παραπέμπει στο δικαστήριο του Λουξεμβούργου διότι πρέπει να διατηρηθεί κατά την άποψή μου το, μονοπόλιο της ερμηνείας της συνθήκης ε, από το δικαστήριο του Λουξεμβούργου. το αν τώρα μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα ακολουθηθεί η διαδικασία του προδικαστικού ερωτήματος που άκουσα σε αυτή τη συζήτηση, αυτό είναι ένα θέμα προς συζήτηση και επίλυση. Τώρα, στο δεύτερο ερώτημα, ως προς τους ε, συμμετέχοντες διαδίκους, ε, ε, νομίζω ότι πρέπει να αναπροσαρμοστούν οι υπάρχουσες διατάξεις της ΕΣΔΑ που επιτρέπουν τη συμμετοχή τρίτου πλην του προσφεύγοντος και του απευθείας ενεγωμένου. Ε, προς το σκοπό να εξασφαλιστεί με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενότητα και ασφάλεια δικαίου. Σημασία έχει δηλαδή να μεθοδευτεί η τοποθέτηση σε θέση διαδίκου, είτε δυνητικά είτε υποχρεωτικά κατά περίπτωση, σε θέση διαδίκου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι συζητήσεις, όπως φάνηκε και εδώ, έχουν διαμορφώσει την ιδιότητα του συνεναγωμένου. Ο καινοτόμος αυτός θεσμός πρέπει να διαμορφωθεί με διατάξεις στη συνθήκη προσχώρησης κατά τρόπο σαφή αλλά και αρκετά ευρύ ώστε να διευκολύνεται ήδη υπάρχουσα καλή συνεργασία μεταξύ των ε, δύο δικαστηρίων. Πιο συγκεκριμένα και όσο γίνεται πιο συνοπτικά η διαμόρφωση της μορφής του συναναγωμένου ε, που δεν ε, έχει ανταπόκριση τουλάχιστον τώρα στις ισχύουσες διατάξεις της ΕΣΔΑ ε, είναι, εμφανίζει αρκετές περιπλοκές στις οποίες όμως μπορεί να δίνεται η παρακατολίση. Όπου προσβάλλεται οποιασδήποτε φύσης πράξη κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνεπάγεται εφαρμογή του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης η πράξη, πράξη οποιασδήποτε μορφής της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή οργάνων της δικαίωμα συνεναγωμένου πρέπει να έχει οπωσδήποτε η Ευρωπαϊκή Ένωση και σε αντίστοιχη περίπτωση βέβαια το κράτος μέλος και αυτά ε, ξεκαθαρίζονται στο σημείο 7 και 8 της έκθεσης με το σωστό τρόπο διότι έτσι μπορεί να αποφευθεί η δημιουργία παρερμηνιών και κενών. Το ερώτημα είναι όμως πώς θα εξασφαλιστεί αυτή η συμμετοχή θα πρέπει να γίνεται γνωστοποίηση της υπόθεσης ή και πρόσκληση του κατά περίπτωση συναναγωμένου από το Δικαστήριο του Στρασβούργου, μια πρόσθετη επιβάρυνση γραφειοκρατική στο σύστημά του, ή θα αφαιθεί το θέμα να ρυθμιστεί με εσωτερικό κείμενο συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών μελών, ένα κείμενο εσωτερικό που νομίζω ότι ούτως ή άλλως πρέπει να διαμορφωθεί και εν ώψη άλλων θεμάτων. Όπως παραδείγματος χάρη πώς θα εκτελεστεί μια καταδίκη από το δικαστήριο του Στρασβούργου χρηματική ή αποκατάστασης αλληλεγγύος ή ολόκληρο ή κατά ποσοστό εναντίον και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του κράτους μέλους, όπως και άλλες περιπτώσεις. Αυτές οι δικαστικές, διαδικαστικές λεπτομέρειες πρέπει να εντοπιστούν και να ρυθμιστούν με γνώμονα αφενός τη μη πρόσθετη επιβάρηση του δικαστηρίου του Στρασβούργου και αφετέρου τη διευκόλυση ύπαρξης διακριτικών ευκαιριών στη σχέση μεταξύ των Ευρωπαϊκής Ένωσης και κρατών ε, μελών. Και τελευταίο ως προς τη σχέση των δύο Ευρωπαϊκών Δικαστηρίων, ε, βεβαίως όπως επισημαίνεται και στο σημείο 1 της έκθεσης, δεν είναι σχέση ιεραρχική, αλλά είναι σχέση εξειδίκευσης, όπως προέκυψε και από τις θέσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης. Το ένα δικαστήριο του Λουξεμβούργου έχει αντικείμενο την ερμηνεία και εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης, ε, η οποία όμως περιορίζεται κατά το σκέλος που πλέον η κρίση επί της ΕΣΔΑ θα μεταφέρεται στο δικαστήριο του Στρασβούργου. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι το Λουξεμβούργο αποξενώνεται από το πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διότι μπορεί να εμπλακεί στου ίδιου είδους υπόθεση από φορμή άλλη ένδικη υπόθεση, αλλά και πάντως παραμένει ακάλυπτος ο χώρος των κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων που καλύπτεται από το χάρτη και όχι από την ΕΣΔΑ. Ε, παρά την υφιστάμενη άριστη συνεργασία των δύο δικαστηρίων και το σεβασμό της Εκατία νομολογίας υπάρχουν ζητήματα που δημιουργεί η νέα κατάσταση η οποία κατά την άποψή μου απαιτεί απευθεία συνεννόηση των δύο δικαστηρίων. Και ε, ακόμα και το θέμα του ελέγχου του πρωτογενούς δικαίου πρέπει να επιληθεί μεταξύ των δύο δικαστηρίων. Ε, αυτά ε, τώρα ως προς τα όργανα της ΕΣΔΑ ο χρόνος ε, συμπληρώθηκε αλλά έχει φάνηκε οριμάσει η ιδέα της συμμετοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης με δικαστή, τη συμμετοχή στην ε, Επιτροπή των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, της, ε, στην Επιτροπή των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης και στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση και είναι θέματα μάλλον τεχνικά που νομίζω ότι μπορούν να ξεκαθαριστούν. Ευχαριστώ πολύ. E Ευχαριστούμε. Ε, είναι δυσάρεστο βέβαια. Είναι δυσάρεστο όταν πιέζω να ε, συντηρηθεί ο χρόνος των ομιλητών. Αλλά ε, ελπίζω να έχουμε και τα γραπτά σας κείμενα. Αφήστε μας πριν φύγετε το κείμενο στη γραμματεία εδώ, η οποία θα φροντίσει να μοιραστούν σε όλους τους ευρωβουλευτές μέλη της Επιτροπής μας ενδεχομένω και με μετάφραση, κάποιο τρόπο, προσπαθήσουμε να μεταφραστούν ορισμένα κείμενα. Και μπαίνουμε στην τελευταία φάση της συνεδρίασης. Δεν ξέρω αν κάποιος θέλει να πάρει το λόγο. Κανείς δεν ζητάει το λόγο. Ας δώσουμε λοιπόν το λόγο στη συνάδελφο Χαουρέγη. Ο Χαουρέγη θα κάνει ερωτήσεις στην τελευταία αυτή φάση. Δεν φτάσαμε ακόμα στο τέλος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω κάποιες ερωτήσεις για τον κύριο Γιάκομς και επίσης και για τον εκπρόσωπο του Συμβουλίου της Ευρώπης. Πρώτα απ' όλα, θεωρείτε εσείς ή θεωρείτε κύριε Γιάκομς ότι θα χρειαζόταν να εξασφαλιστεί η παρουσία ενός Ευρωπαίου δικαστή στην διαδικασία εξέτασης του δικαστηρίου του ΕΔΑΔ για περιπτώσεις που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι θέμα οργάνωση εσωτερική του δικαστηρίου. Ίσως η κυρία δικαστή μπορεί να απαντήσει στο θέμα αυτό, γιατί φυσιολογικά συμμετέχει ο δικαστή κάθε κράτου διάδικου όταν πρόκειται για ένα θέμα που αφορά αυτό το κράτο. Αυτό κατά τρόπον ώστε να μπει στο σωστό πλαίσιο η νομική πράξη, ο νόμος ο οποίος διαμφισβητείται. Δεν έχει τελική συμμετοχή στην απόφαση. Το ερώτημα είναι αν οι εσωτερικοί κανόνες που ισχύουν στο ΕΔΑΔ μας εξασφαλίζουν ότι ο Ευρωπαίος δικαστής θα έχει τη δυνατότητα να είναι πάντα παρόν σε οποιαδήποτε περίπτωση που χρειάζονται να δοθούν εξηγήσει και το σωστό πλαίσιο σε σχέση με ένα νομοθέτημα ευρωπαϊκού δικαίου. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα που θα σας θέσω. Το δεύτερο ερώτημα. Υπάρχει μια σειρά φορέων που δεν ξέρω αν πράγματι είναι τμήμα της σύμβασης ή δεν ξέρω ακριβώς ποια είναι η δυνατότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση να συμμετάσχει σε αυτούς τους φορείς μέσω της Κομισιόν με καθεστώς παρατηρητή ή οτιδήποτε άλλο στους εξής φορείς. Στον εκπρόσωπο, στον Επίτροπο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων, στην Διακυβερνητική Επιτροπή για τις Μεταναστεύσεις της, του Συμβουλίου της Ευρώπης, στον Φορέα για την ε, προστασία από την, ε, τους βασανισμούς ή τις απάνθρωπες και εξευθυλιστικές μεταχειρήσεις. Θέτω αυτό το ερώτημα γιατί υπήρξε μια τροπολογία από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων που ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διεκδικήσει την παρουσία παρατηρητού από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα θέματα αυτά. Θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η νομική χρειά αυτών των φορέων και μέχρι ποιου σημείου η παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην, ως, ως ε, συμβαλόμενου μέρους στην σύμβαση προκαλεί κάποια αποτέλεσμα σε σχέση με την παρουσία τους αυτούς τους φορείς. Τρίτον, θα ήθελα να επανέλθω στο ότι η επιχειρηματολογία για την μη ύπαρξη προσφυγών μεταξύ κρατών μελών δεν προκύπτει μόνο από το άρθρο 344 για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά συγχρόνως και, στο άρθρο, και από το άρθρο 55 της ίδιας της σύμβασης <clears throat> που θεσπίζει μια συμφωνία μεταξύ των συμβαλωμένων κρατών να μην χρησιμοποιήσουν τη σύμβαση ώστε να προσφύγουν κατά ενός άλλου συμβαλόμενου μέρους, ενός άλλου συμβαλόμενου κράτους. Το λέω αυτό γιατί η εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύει τα κράτη-μέλη της να μην έχουν αμοιβέ μεταξύ τους ε, προσφυγές έχει διπλή βάση, όχι μόνο το 344, αλλά και το 55 της Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Αυτά είναι τα ερωτήματά μου. Ευχαριστώ. Yes, uh, uh Ευχαριστώ. Ίσως η ερώτησή μου να είναι αφιλής. Ο καθηγητή Τζέκομ είπε ότι το δικαστήριο της Στρασβουργού θα έχει ουσίες να ακυρώσει την νομοθεσία της Ένωσης. Το ξέρουμε αυτό, αλλά δεν ξέρουμε, τουλάχιστον εγώ δεν ξέρω, ότι θα έχει κάνει την εξουσία να δηλώσει την νομοθεσία ασύμβατη με την ε, ΕΣΔΑ. Φαντάζομαι ότι θα χρειάζεται όχι απλώς να δράσουμε σε σχέση ε, μία απάντηση είναι ασύμβατη νομοθεσία. θα πρέπει να περιμένουμε η νομοθεσία να αρχίσει να ισχύει και μετά η συμπεριφορά του πώς θα ισχύει να τεθεί ένα αμφιβόλο και όχι η νομοθεσία πάνω στην οποία στηρίχτηκε. Βέβαια, η μόνη αναφορά στον νόμο θα, γίνει, θα είναι στην ΕΣΔΑ και όχι στην νομοθεσία της Ένωσης ή την εθνική νομοθεσία κράτους μέλους που οδήγησε στη συγκεκριμένη συμπεριφορά δεν ξέρω αν η ερώτησή μου ήταν σαφής. Πάντως αυτή ήταν η ερώτησή μου. Πρόεδρος, ας αρχίσουμε τις απαντήσεις. Ο συνάδελφος με τις ερωτήσεις του συναδέλφου Χαρική. Οι εμπειρογνώμονες ποιος θέλει. Ο κύριος Γιάκοψη, η, η κυρία Τούλκενς, ποιος θέλει πρώτος. Ah. Συγγνώμη, νομίζω ότι το πρώτο ερώτημα, αν τα πάρω τα ερωτήματα με τη σειρά τους, για το ρόλο του δικαστή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν θα πρέπει να παρήσατε σε όλες τις περιπτώσεις όπου εμπλέκεται το ευρωπαϊκό δίκαιο, νομίζω ότι αυτή την ερώτηση πρέπει να την απαντήσει η κυρία Τούλκενς που ξέρει πολύ καλύτερα το σύστημα. Ίσως μπορώ να επανέλθω στα άλλα ερωτήματα εγώ. Δε μεγάλη χαρά λέει η κυρία Τούλκενς διότι πάντα ο εθνικός μεσαισαγωγικά δικαστής προβλέπεται να είναι παρόν στη διαδικασία όλων των υποθέσεων που εμπλέκουν τη χώρα του. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία, αυτό σημαίνει ότι έχει τη δυνατότητα να ψηφίζει για όλες τις περιπτώσεις που αφορούν τη χώρα του, όχι μονάχα στα τμήματα, αλλά και στην, στο ανώτατο όργανο του ΕΔΑΔ. Το λέει εκπεφρασμένα λοιπόν η σύμβαση ότι ο κάθε δικαστής λειτουργεί μεμονωμένα, ότι ο, ρόλος ενός δικαστή δεν είναι προφανώς να υπερασπιστεί τη χώρα του και τα θεσμικά όργανα της χώρας του, αλλά να εξηγήσει τις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά που μπορεί να έχει το εθνικό δίκαιο. Αυτό είναι ουσιαστικό λοιπόν θέμα. Σε ό,τι αφορά επομένω ένα δικαστή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να έχει ακριβώ το ίδιο καθεστώ όπω και οι άλλοι δικαστέ. Νομίζω ότι αυτή θα ήταν η προτιμητέα ε, λύση, να έχει το ίδιο καθεστώς με τους άλλους δικαστές, να είναι συνυπεύθυνος φυσικά με τους άλλους δικαστές που προέρχονται από τα 47 κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά την ερμηνεία της Σύμβασης Ανθρωπινών Δικαιωμάτων. Φυσικά αυτό μπορεί να τύχει συζήτηση. Μπορεί να πει κάποιο γιατί θα έπρεπε να έχει υποδέστερη θέση ο δικαστής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί στις περιπτώσεις που δεν εμπλέκουν το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχει μόνο ένα συμβουλευτικό χαρακτήρα. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να το συζητήσει κανείς. Εγώ, η δική μου προτίμηση, η προσωπική είναι να συμμετέχει και σε διαβουλευτικό και σε ουσιαστικό επίπεδο δικαστής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί η ιδέα των δικαστών είναι να εξασφαλίζουν συλλογικά την εφαρμογή του δικαίου στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Όλες οι χώρες λοιπόν αυτές που έχουν ε, συνυπογράψει τη Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 47 χώρε και τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση συλλογικά συμμετέχουν στην εξασφάλιση του δικαίου. Αυτό μου φαίνεται ότι είναι μια πολύ ισχυρή αρχή η οποία πρέπει να συνεχίσει να την χάνει σεβασμού. Αυτό είναι για το πρώτο σα ερώτημα. Και θα επανέλθω μετά στο ερώτημα μετά από τον κύριο Γιάκοψ όμω. Um, um, σας ευχαριστώ να πω πώς είναι δική μου άποψη. Η λύση που θα πρέπει να ακολουθηθεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση ως μέλος της σύμβασης είναι ότι το σύστημα θα πρέπει να εφαρμοστεί κατά το δυνατόν όσο πιο πλήρως γίνεται. Σε ό,τι αφορά το ρόλο του δικαστή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να απαντήσουμε και τα άλλα ερωτήματα εν συντομία. Το επόμενο ερώτημα ήταν για την εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε άλλες επιτροπές του Συμβουλίου της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένης της Επιτροπής κατά το βασανιστήριων και τα κοινωνικά δικαιώματα και το καθεξής. Η αρχική μου απάντηση θα ήταν ότι δεν έχω την εντύπωση ότι η συμμετοχή στα σώματα αυτά θα ήταν απαραίτητη απόρρια της προσχώρησης της Ένωσης στην ΕΣΔΑ. Φυσικά γνωρίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι, συμμετέχει ήδη σε πολλές συμφωνίες του Συμβουλίου της Ευρώπης και στο έργο των ε, σχετικών οργάνων, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει απαραίτητα σύνδεση με την ε, Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Για το επόμενο ερώτημα, για το άρθρο 55 της ε, ΕΣΔΑ και την δυνατότητα διακρατικής εφαρμογής. Έχω την εντύπωση ότι πρόκειται για έναν τομέα όπου η προσχώρηση της Ένωσης προκαλεί κάποια ειδικά προβλήματα, γιατί αφενός ε, πρέπει και τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση να συμμετέχουν στις διαδικασίες στο δικαστήριο, αν υπάρχει πιθανότητα να συμπεριληφθεί μέτρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφετέρου μπορεί να υπάρχουν λόγοι για να εξαιρεθούν δράσεις ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα πρέπει να ληφθούν υπόψη κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και θεωρώ ότι θα πρέπει να τραποποιηθεί κάπως το σύστημα της ε, σύμβασης, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να επιληθούν με άμεσο τρόπο, με, για παράδειγμα, τροποποίηση του κανονισμού σε ό,τι αφορά το δικαστήριο αφενός και συμφωνίες αφετέρου μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα δεν θα χρειαστεί απαραίτητα τροποποίηση της ίδιας της σύμβασης. Και φυσικά θα ήταν προτιμητέο να ακολουθηθεί μια διαδικασία τέτοια. Για την τελευταία τώρα ερώτηση ω προ την απόφαση του Δικαστηρίου του Στρασβούργου για τη συμβατότητα των μέτρων τη Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Σύμβαση. Η θέση είναι η εξή. Σε μια φυσιολογική περίπτωση ατομική προσφυγή, τα άτομα τα οποία ε, προσφεύγουν για παραβίαση δικαιωμάτων ε, στο δικαστήριο των ανθρώπινων δικαιωμάτων, αν αποφανθεί ότι υπάρχει όντως ε, παραβίαση, μπορεί η νομοθεσία, αυτό δεν σημαίνει ότι η νομοθεσία είναι απαραίτητα σύμβατη, μπορεί να είναι ο τρόπος εφαρμογής της νομοθεσίας, ο ήταν σύμβατο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κληθεί να αποφασίσει πώς θα αντιμετωπίσει αυτή την παραβίαση και ενδεχομένως να προβεί σε τροποποίηση της νομοθεσίας διαφέρουν τα πράγματα στις ε, περιπτώσεις μεταξύ κρατών, γιατί εκεί τίθεται θέμα σύμβασης με την συνθήκη, με τη σύμβαση γενικά. Δεν πρόκειται για θύματα μεμονωμένα πλέον. Η κατάσταση λοιπόν θα είναι πολύ ιδιαίτερη και αυτό φυσικά ε, θα αποτελεί μια μεγάλη εξαίρεση. Δεν υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα στο Στρασβούργο. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν υπήρξαν τέτοιες περιπτώσεις, αλλά τουλάχιστον σε μια μεγάλη πλειονότητα το Δικαστήριο των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων δεν ασχολείται με τη συμβατότητα μέτρων με τη σύμβαση, μόνο με τον τρόπο εφαρμογής της νομοθεσίας, ο οποίος ενδεχομένως προκάλεσε παραβίαση δικαιωμάτων. Ευχαριστώ. Κύριε Τούρκινς, θα ήθελα να συνεχίσει λίγο στο θέμα αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε δύο πράγματα. Από τη μια μεριά, γιατί έγινε η προσφυγή και ποια είναι η σημασία των αποφάσεων στην αρχή, και αυτό είναι το αλφαβήτα της λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, έχουμε μια περίπτωση εφαρμογής. Υπάρχει μια προσφυγή, ένα παρά κάποια διαμαρτυρία από ένα άτομο κλπ. που ισχυρίζεται ότι είναι θύμα μια παράβασης της νομοθεσίας. Και είναι σημαντικό αυτό, γιατί ο ρόλος μας δεν είναι να μελετήσουμε γενικά, είναι abstracto το κατά πόσο συμφωνεί όχι μια εθνική νομοθεσία με την σύμβαση, η συγκεκριμένη εφαρμογή της συγκεκριμένη περίπτωση για ένα άτομο, για μια ομάδα που ισχυρίζεται ότι υπήρξαν θύμα της παραβίασης αυτής, παράβασης αυτής μάλλον. Γιατί δεν θα είχε καμία νομιμότητα να μελετήσει να αυστράκτω την νομοθεσία γενικά. Μέσα μια συγκεκριμένη περίπτωση πάντα γίνεται αυτό. Το ίδιο και για την Ένωση. Είτε πρόκειται για μια πράξη της Ένωσης ή για μια εθνική πράξη που εφαρμόζει όμως μια πράξη της Ένωσης. Και με την απόφαση θα διαπιστωθεί αν υπήρξε παράβαση της ε, σύμβασης. Η σύμβαση προβλέπει τα κράτη-μέλη να σέβονται τις αποφάσεις του δικαστηρίου και όλο και περισσότερο σήμερα λέμε αν μια απόφαση του δικαστηρίου αφορά μια χώρα θα πρέπει και οι άλλες χώρες να εμπνέονται από τις κατευθυντήριες γραμμές για να αλλάξουν την νομοθεσία τους. Μετά γίνεται αυτό. Άρα οι αποφάσει τι λένε. Πρέπει να αλλάξουν αυτό που δημιούργησε το πρόβλημα, το συγκεκριμένο πρόβλημα. Δεν θα ακυρωθεί μια νομοθεσία. Δεν θα ακυρώσουμε μια δίκη. Όχι. Θα πούμε σε ένα κράτο υπήρξε παράβαση. Στο σημείο αυτό εσείς υπό τον έλεγχο του Συμβουλίου Υπουργών να γίνει η αλλαγή in Αυτή είναι η ισχύς και ο περιορισμός της προσχώρησης στην ε, σύμβαση. Και από την άλλη μεριά το τι γίνεται με την εκτέλεση των αποφάσεων. Κύριε Πρέσβη, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πάρα πολύ σύντομα απλώς να απαντήσω στο συγκεκριμένο αυτό ερώτημα, το οποίο νομίζω ότι απευθύνθηκε σε μένα από τον κύριο Χαουρεγή. Πρώτα απ' όλα μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι σε ό,τι αφορά την ε, διακυβερνητική διευθύνουσα επιτροπή στο Συμβούλιο της Ευρώπης, προβλέπεται η πρόσκληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με καθεστώς παρατηρητή όπως και στην Επιτροπή Ανθρωπινών Δικαιωμάτων και στην ε, Κατευθύνουσα Επιτροπή για τα θέματα μετανάστευσης για τα περαιτέρω βήματα τα οποία μπορούσαν να ληφθούν για να συμπληρωθεί η προσχώρηση Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στον τομέα της συνεργασίας για τα θεμελιώδη δικαιώματα. Το Συμβούλιο της Ευρώπης με μεγάλη ικανοποίηση καταγράφει αυτή τη σύσταση που περιλαμβάνεται στην έκθεσή σας, στο ψηφισμά σας σε σχέση με την ενδεχόμενη προσχώρηση στην κοινωνική στη χάρτα του 1961 και την αναθεωρημένη μορφή της του 1976 και αναφερθήκατε και στην πρόταση τροπολογίας της Επιτροπής Εξωτερικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η οποία ζητά να υπάρξει παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη συνεργασία με ειδικευμένους φορείς του Συμβουλίου της Ευρώπης. Εδώ θα ήθελα να καλωσορίσω αυτή την τόσο ενδιαφέρουσα πρόταση και να αναφέρω ότι το θέμα αυτό θα μπορούσε να εξεταστεί και για άλλα σώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως είναι το Συμπητή Φορέας για την πρόληψη της, ε, τον... του βασανισμού, τον φορέα κατά του ρατσισμού και της μυσαλλοδοξίας και τον φορέα για την αποτελεσματικότητα της απόδοσης δικαιοσύνης. Τέλος κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας αναφέρω ότι στις 24 καθώς και τις 25 Μαρτίου ο Διευθυντή του Συμβουλίου της Ευρώπης για την παρακολούθηση αυτών των θεμάτων θα είναι παρόν στις Βρυξέλλες για να έχει επαφές με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα χαρώ ιδιαίτερα να διευκολύνω, ενδεχομένως εάν σας ενδιαφέρει, μια διμερή συνάντηση του εισηγητού με τον αρμόδιο διευθυντή όταν θα είναι εδώ την επόμενη εβδομάδα. Το σημειώνει αυτό ο ηγητής, φαντάζομαι, τη συνάντηση αυτή. Δεν ξέρω αν η κυρία Μπενάκη θα ήθελε να προσθέσει κάτι, αν θέλει. Όχι. Τότε ας δώσουμε το λόγο στον εισηγητή μας για τα πρώτα συμπεράσματα αυτή την, από την πολύ αυτή πλούσια συνάντηση, η οποία απλοποίησε ορισμένα θέματα, περιέπλεξε άλλα, πάντως ήταν πάρα πολύ χρήσιμη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι, κυρίε και κύριοι, Δυστυχώ πρέπει κάποια στιγμή να κλείσουμε αυτή τη τόσο πλούσια, όπω είπε ο Πρόεδρος, και ενδιαφέρουσα συνάντηση. Δεν πρόκειται να σας ταλαιπωρήσω με συμπεράσματα τα οποία ήδη τα έχετε αντλήσει όλοι από αυτή την συνεδρίαση. Τη στιγμή που βρισκόμαστε προς το τέλος της ημέρας, ούτε είμαι τόσο ανόητος, ώστε να προσπαθήσω να αντλήσω συμπεράσματα στη θέση των ίδιων των εμπειρογνωμόνων. Μόνο οι εμπειρογνώμονες μπορούν να παρουσιάσουν πραγματικά συμπεράσματα. Παρ' όλα αυτά θέλω να πω δύο πράγματα που νομίζω ότι σε πολιτικό επίπεδο θα πρέπει να τα τονίσουμε. <clears throat> Γιατί το νομικό πλαίσιο, το νομικό, ο νομικός χαρακτήρας αυτής της συνεδρίασης δεν μας επέτρεψε να υπενθυμίσουμε ότι καταρχήν με την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ΕΣΔΑ περατώνεται μία μακ... μακροσκελής διαδικασία διεκδικήσεων που συνάπτεται με την ουσία του ευρωπαϊκού εγχειρήματο. Ότι δηλαδή η έννοια αυτή, <clears throat> η αντίληψη που είχε η Ευρώπη πάντα, ότι το άτομο και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τα θεμελιώδη του δικαιώματα και οι ελευθερίες του, το κράτος δικαίου, η δημοκρατία είναι πάντα στο κέντρο του ευρωπαϊκού εγχειρήματο, έτσι πραγματώνεται γιατί πέραν από γεωστρατηγικές αναγκαιότητες, οικονομικές κατασκευές ενό κοινού χώρου εσωτερικής αγοράς και όλα αυτά, ή τουλάχιστον παράλληλα με όλα αυτά, νομίζω ότι είναι απαράγραπτο να μην ξεχάσουμε και να τονίσουμε ότι στην απαρχή της ευρωπαϊκής ιδέας υπάρχει αυτό το εγχείρημα εκπολιτισμού, το να υπάρξει αυτό το σύμβολο της ευρωπαϊκής ταυτότητα, το οποίο με την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με την προσυπογραφή της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ουσιαστικά πραγματών αυτήν την τόσο παλιά διεκδίκηση του, των πατέρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμα και του ίδιου του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και είναι απόρρια και κατάληξη όλου αυτού του ευρωπαϊκού κινήματος για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ήταν πολύ πλούσια αυτή η διαδικασία, η οποία απολύγει επιτέλους τη δυνατότητα να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση ένα αρμονικό ένομο πλαίσιο και το οποίο περιλαμβάνει τις απαραίτητες διαφυλάξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Όμως πρέπει να υπενθυμίσω ότι το πολιτικό σύστημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή ή μέχρι αυτή τη στιγμή έχει προωθηθεί από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θέτω αυτό το ερώτημα και νομίζω ότι κάθε ένας μας έχει το δικαίωμα να θέσει αυτό το ερώτημα μέχρι ποιου σημείου τα κράτη-μέλη και γνωρίζω ότι η προσχώρηση της ΕΣΔΑ είναι εντολή τη συνθήκη Λισαβόνα. Επομένω, ήταν μια απόφαση που ελήφθη από τα ίδια τα κράτη-μέλη. Αναρωτιέμαι σε ποιο βαθμό τα κράτη-μέλη θέλουν πράγματι να προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Θα πρέπει να έχουμε επίγνωση του γεγονότο ότι στην ευρωπαϊκή πολιτική συζήτηση αυτή τη στιγμή είναι άλλα θέματα τα οποία έχουν προτεραιότητα. Καταρχήν η τεράστια αυτή ανάγκη να δοθούν απαντήσεις στην οικονομική κρίση και πολλά κράτη-μέλη βλέπουν αυτή τη διαδικασία προσχώρησης ως μια πρόσθετη επιπλοκή ή περιπλοκή, σαν προσθήκη ενός ακόμα δικαστηρίου στην ένωμη τάξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μπορεί να υποβάλει σε εξωτερικό έλεγχο τις αποφάσεις και τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πράξεις που αποτελούν αντικείμενο κοπιωδών διαπραγματεύσεων σε καθημερινό επίπεδο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό θέλω να τονίσω, κύριε Πρόεδρε, ότι και σε αυτή την περίπτωση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να παίξει το σημαντικό ρόλο κινητήριου μοχλού και αυτού ο οποίος παροτρύνει και προωθεί μια απόφαση η οποία μπορεί να έχει ληφθεί βέβαια σε επίπεδο συνθήκης αλλά όπως υπενθυμίσαμε, θα, απο, θα απαιτήσει και μια πολιτική προσπάθεια για να εφαρμοστεί στην πράξη. Δεν λέω ότι υπάρχει αντίθετη αντιμετώπιση από κάποια κράτη-μέλη. Λέω απλώς ότι υπάρχει ίσως κάποια αδιαφορία σε σχέση με αυτή την προσχώρηση. θα φανεί ενδεχομένως και από την ίδια τη διαπραγμάτευση. Πρέπει ακόμα να διασαφηνίσουμε ποιο είναι το περιεχόμενο αυτής της διαπραγμάτευσης για την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ΕΣΤΑ και βλέπουμε ήδη ότι η Κομισιόν φυσιολογικά θα πρέπει να είναι αυτή που θα αυτοπεριοριστεί κατά κάποιο τρόπο μέσα στα πλαίσια αυτής της διαπραγμάτευσης. Προφανώς είναι γεγονός ότι η Κομισιόν έχει διεκδικήσει το αποκλειστικό δικαίωμα διαπραγμάτευσης. Είναι ένα δικαίωμα το οποίο έχει αλλά ήδη έχει θεσπίσει ορισμένα όρια λέγοντας ότι μέσα στα πλαίσια αυτής της διαπραγμάτευσης μόνο η Κομισιό θα διαπραγματευτεί και συγχρόνως ζήτησε από τα κράτη-μέλη <clears throat> να λειτουργήσουν σε αρμονία με αυτά τα οποία θα διαπραγματευτεί η Κομισιόν εκπροσωπώντας όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Είναι λογικό λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να πληροφορήσει τα κράτη-μέλη ότι τα 27 αυτά κράτη που είναι τμήμα των 47 μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης θα πρέπει να παραμείνουν πιστά στις θέσεις τις οποίες εκφράζει η Κομισιόν, αλλά η Κομισιόν στη χθεσινή τη συμφωνία μας προειδοποίησε ότι θα συνοδεύεται αυτή η προσχώρηση από διατύπωση επιφυλάξεων και από συγκεκριμένες δηλώσεις. Αυτό δεν μπορώ να πω ότι με βασανίζει ακόμα, αλλά με ανησυχεί. Γιατί αρχίζει να διαφαίνεται η δυνατότητα <clears throat> και το ενδεχόμενο η Κομισιόν να θωρακίζεται με την δημιουργία, με τη διατύπωση επιφυλάξεων που θα προκύψουν από ορισμένα κράτη-μέλη. Εγώ τονίζω και πάλι ότι δεν μπορούμε να επηρεάσουμε τις αρμοδιότητες και τις εξουσίες και αυτό είναι και, το, και η εντολή που έχει προκύψει σε σχέση με τη διαπραγμάτευση αλλά θα πρέπει να θεσπίσουμε, να έχουμε και μια θέση ενώπιον των πρωτοκόλων που συνοδεύουν τη σύμβαση ΕΣΔΑ η Κομισιόν που είναι ίσως ευφυής αλλά δεν ακολουθούν τη γραμμή που ανέφερε το αρχικό εγχείρημα και την αρχική πολιτική θέληση, όπως είπε και ο κ. Ζακέ. Η ιδέα αυτή της κυρίας Ρέντιν, ότι πρέπει να αναγνωριστεί το δικαίωμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να, προσχωρεί, να προσχωρήσει στη σύμβαση και σε οποιοδήποτε από τα πρωτόκολλα της σύμβασης τώρα ή στο μέλλον, αυτό προαναγγέλει Κάτι με το οποίο δεν μπορούμε να είμαστε ίσως όλοι σύμφωνοι. Η Κομισιόν προσπαθεί με ένα σόφρονα και προσεκτικό τρόπο να βρει μια μορφή ε, προσχώσεις μόνο στα πρωτόκολλα τα οποία έχουν υπογράψει όλα τα κράτη-μέλη και αφήνει ανοιχτό το μέλλον για μια μεταγενέστερη προσυπογραφή ad calendas grecas όπως είπε ο Ζαλ Πολ στο Δινεκές για τα υπόλοιπα πρωτόκολλα. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρόβλημα το οποίο μπορεί να προκύψει ενώπιόν μας και να φανεί πολύ σημαντικό στη διαδικασία αυτή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ζητήσει μέσω της ε, εντολής της Κομισιόν από ό,τι προβλέπουμε να υπάρχει και μια παρουσία μεταξύ των δικαστών, παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης μεταξύ της Επιτροπής Υπουργών με δικαίωμα ψήφου, γιατί αυτή είναι η πρόταση την οποία έχει διατύπωση η Κομισιόν, και επίσης τη συμμετοχή στην κοινοβουλευτική συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπη παρά το γεγονός ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μου φαίνεται κάπως αυτή η συμμετοχή μου φαίνεται λιγάκι περίτη. Σε τελική ανάλυση και εν τέλει όπως ελέγχθη εδώ διάφορες φορές η Κομισιόν θα πρέπει να διεκδικήσει τον χαρακτήρα της συνεναγόμενες σε θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορεί κανείς να έχει τη δική του άποψη για τα στοιχεία που θα προκύψουν από αυτό και επίσης η Κομισιόν θα προσπαθήσει, φαντάζομαι, να προχωρήσει σε μια επισημοποίηση της δέσμευσης των κρατών μελών να μην έχουν αμοιβέ μεταξύ τους και εναντίον τους προσφυγές. Κλείνω με μια τελευταία παρατήρηση. Αυτή τη στιγμή το επόμενο βήμα που πρέπει να κάνουμε στους επόμενους μήνες είναι ακριβώς να υπάρξει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η έκθεση την οποία εκπονεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα είναι ένα έγγραφο πολύ πιο πλούσιο από αυτό που έχετε δει μέχρι στιγμής γιατί ακόμα οι διάφορε κοινοβουλευτικέ ομάδες και οι διάφορε κοινοβουλευτικέ επιτροπές θα πρέπει να προσθέσουν τι δικές τους προτάσεις και να συμβάλλουν στην εκπόνηση μιας τελικής έκθεσης Και εγώ πιστεύω, αν δεν με διορθώσει ο πρόεδρος Κασίνη, ότι κατά πάσα πιθανότητα τον Ιούνιο, το αργότερο, θα μπορέσει να εγκριθεί από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αυτή η έκθεση. Συγχρόνως όμως είναι παράλληλο, είναι απαραίτητο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να εγκρίνει ομόφωνα την εντολή διαπραγμάτευσης της Κομισιόν. Και εδώ ανοίγω μια παρένθεση σε σχέση με την θέση των κρατών μελών. Γιατί ευτυχώ η Κομισιόν έχει κάνει τα απαραίτητα, αλλά τώρα πρέπει το Συμβούλιο και με ομοφωνία να εγκρίνει τη διαπραγματευτική εντολή της Κομισιόν και ελπίζουμε λοιπόν, αν θέλει ο Θεός, να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις πριν από το καλοκαίρι, τον Ιούνιο, έστω τον Ιούλιο, να γίνει αυτό δυνατό. Ελπίζουμε, γιατί θα πρόκειται για διαπραγματεύσεις που θα κρατήσουν κάποιους μήνες και που στη συνέχεια θα επιτρέψουν μια τρίπλη διαδικασία, την οποία και αυτή θέλω να σας υπενθυμίσω. Δηλαδή, πρώτον, ότι θα υπάρξει έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο της διαπραγμάτευσης, των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης. Δεύτερον, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πρέπει και αυτό να εγκρίνει ομόφωνα αυτή τη συμφωνία που θα γίνει και τρίτον θα πρέπει να υπάρξει βάση των συνταγματικών διατάξεων κάθε κράτους μέλους η κύρωση από όλα τα κράτη-μέλη. Ξέρετε ότι αυτή η κύρωση, κύρωση οδηγεί σε εκπλήξεις, σε ανησυχίες και σίγουρα είναι μια χρονοβόρα διαδικασία. Όλα αυτά μας κάνουν να πιστεύουμε ότι αν πάνε όλα καλά, ίσως το τέλος του έτους 2011 να έχει γίνει πραγματικότητα η προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μακάρι. Και σας ευχαριστώ κυρίες και κύριοι. Ε, Επομένω μπορούμε να κλείσουμε την σημερινή συνεδρίαση. Ευχαριστώ και πάλι του καθηγητέ, του ακαδημαϊκού, του πανεπιστημιακού, του εκπροσώπου Συμβουλίου τη Ευρώπη, του δικαστέ, όλου του παρόντε για τη συμμετοχή σας, πάρα πολύ σημαντική. Εμείς από τη μεριά μας ως Επιτροπή έχουμε ορίσει 25 Μαρτίου ημερομηνία για τροπολογίες στο κείμενο Χάργη. Επιβεβαιώνεται η ημερομηνία για τροπολογίες 25 Μαρτίου. Η συζήτηση θα γίνει μετά στις 6 Απριλίου. Ενδεχομένω το Μάιο η ψηφοφορία. 6 Απριλίου, επαναλαμβάνω, θα συζητηθούν τροπολογίες ψηφοφορία το, το Μάιο, Ολομέλεια Ιουνίου. Αυτό είναι το πρόγραμμά μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Arrivederci.